Oh, Good morning. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή συνεδρία. Ως πρώτη της Επιτροπής ΙΜΚΟ θα ήθελα να καλωσορίσω ε, την προτινόμενη Επίτροπο Σιλβί Γκουλάρ για την δεύτερη ακρόασή της, κάτι που ζήτησαν οι συντονιστές της Επιτροπής ΙΜΚΟ και ΙΤΡΕ. Να καλωσορίσω την κυρία Βαγιόν, η οποία είναι υπεύθυνη, είναι μάλλον πρόεδρος της Επιτροπής Ήτρε και από κοινού θα προεδρεύσουμε και βεβαίως τα μέλη των Επιτροπών Ίμκο και Ήτρε που έχουν οργανώσει από κοινού αυτή την ακρόαση. Θέλω να ευχαριστήσω τους προσώπους των Επιτροπών Γιούρι και Κούλτ επίσης που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και από την Επιτροπή Τραν και Σέντε που είναι προσκεκλημένοι. Γνωρίζουμε όλοι γιατί βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Για να υπάρξει περαιτέρω διευκρίνηση στις απαντήσεις που δόθηκαν στην υποψήφια επίτροπο για τα θέματα που ετέθησαν στην πρώτη ακρόαση και κατόπιν υποβλήθηκαν και γραπτά και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό για την Ήτρε το χαρτοφυλάκιο της κυρίας Γκουλάρ γιατί η ψηφιακή ενιαία αγορά είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε από κοινού με την Επιτροπή ε, ε Ήτρε, συγγνώμη, από πλευρά ΙΜΚΟ είναι σημαντική για μένα. Να δώσω το λόγο στην κυρία Βαλέαν. Ευχαριστώ κυρία Ντεσούτερ για την ε, εισαγωγική σας παρουσίαση. Καλώς ορίζω όλους τους συναδέλφους ε, στην συνεδρίασή μας σήμερα και καλώς ορίζω και την υποψήφια επίτροπο κυρία Σιλβί Γκουλάρ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. και καλωσορίζω όλους τους συναδέλφους από τις διάφορες επιτροπές και όσους μας παρακολουθούν μέσω του ίντερνετ. Να σας εξηγήσω πώς θα διεξαχθεί η ακρόαση σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τις καθεντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κοινοβούλιο αξιολογεί τους επιτρόπους, υποψήφιους επιτρόπους στη βάση της Γενικής ε, των γενικών προσόντων του, δέσμευση για την Ευρώπη και προσωπική ανεξαρτησία. Επίση, ε, αξιολογεί τη γνώση του προτινόμενου χαρτοφυλακίου και τι επικοινωνιακέ του δεξιότητε. Πριν από την ακρόαση, η Επίτροπο απάντησε γραπτό σε μια σειρά από συμπληρωματικέ γραπτέ ερωτήσει που έθεσαν τα μέλη ΙΜΚΟ, ΙΤΡΕ, ΚΑΛΤ και Τζούρι. Οι γραπτέ απαντήσει, ΚΑΛΤ και Τζούρι είναι συνδεδεμένε με την Επιτροπή. Οι γραπτέ απαντήσει έχουν διανεμηθεί στα μέλη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκουλάρ για τις απαντήσεις σας στις συμπληρωματικές ερωτήσεις. Για σήμερα. Θα ξεκινήσει η υποψήφια επίτροπης κυρία Γκουλάρ μέχρι 10 λεπτά και μετά θα έχουμε 13 ερωτήσεις από συναδέλφους. Πρώτα εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, 7 ερωτήσεις και οι υπόλοιπε ερωτήσεις μέλη, από μέλη των επιτροπών που συμμετέχουν στην ακρόαση. Κάθε ερώτηση θα είναι 5 λεπτά, μία, ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση, ένα λεπτό για την συμπληρωματική ερώτηση και ένα λεπτό για την απάντηση στη συμπληρωματική ερώτηση. Θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε όσο αυστηρά γίνεται το χρόνο. Κάνω έκκληση να τηρήσετε όλο το χρόνο σας. Αυτά. Κυρία Κουλά, έχετε το λόγο. Δέκα λεπτά παρακαλώ. Κυρίες Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και για όλους όσους μας ακούν εξ αποστάσεως, καλημέρα σας. Μετά από την πρώτη μου ακρόαση στις 2 Οκτωβρίου, ε, μου είπατε ότι θέλετε να απαντήσω σε γραπτές ερωτήσεις, ε, κάτι που έκανε ευχαρίστω γιατί σέβαμε βαθιά το ρόλο του Κοινοβουλίου σε, αυτήν την, ε, σε αυτό το εγχείρημα δημοκρατικών ελέγχων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα είμαι ενώπιον για να εμβαθύνω σωσμένα σημεία. Θέσατε μία νομότυπη ερώτηση γιατί ένα χαρτοφυλάκιο τόσο περίπλοκο, τόσο εκτεταμένο. Πρώτα απ' όλα είναι η στρατηγική επιλογή της ε, Προέδρου, Φοντε Λάιεν, την οποία συμμερίζομαι πλήρως, γιατί νομίζω ότι σωστά αντιλαμβάνεται την περιπλοκότητα των οικονομικών, βιομηχανικών και ανθρωπίνων διακυβευμάτων ε, τα οποία αντιμετωπίζουμε. Έχει έννοια ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο, πρώτα απ' όλα, γιατί οι τεχνολογικές εξελίξεις στην ουσία έχουν καταργήσει τη διαφορά μεταξύ μια ενιαίας αγορά και μια ψηφιακή ενιαίας αγοράς. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των ε, βιομηχανικών προκλήσεων και των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή οικονομία. Όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε είναι να εξυγχρονίσουμε το σύνολο τη οικονομία μα. Παραδείγματα για να είμαι πιο συγκεκριμένοι. Πρώτα απ' όλα, για την βιομηχανία μα, Ξέρετε ότι θέλουμε να έχουμε μια βιομηχανική στρατηγική. Θέλουμε να έχουμε αλυσίδε αξίε που να διασφαλίσουν την τεχνολογική μας κυριαρχία. Να μην υπολοιπόμεθα άλλων ε, περιοχών του κόσμου. Γι' αυτό θα θέλαμε να έχουμε από κοινού και ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους για να αναπτύξουμε νέα προϊόντα, να δημιουργήσουμε νέες αγορές μέσω βιομηχανιών που να καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια ε, ενώ θα παραμένουν ανταγωνιστικές. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τεχνολογίες τομής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Δεύτερον, ένα στόχος της νέας επιτροπής που είναι επίσης ιδιαίτερα φιλόδοξος είναι να περάσουμε για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή στην ε, εξάλληψη της χρήσης άνθρακα. Και ε, με κακή τεχνική ορολογία θέλουμε να έχουμε επίσης την κυκλική οικονομία. Δηλαδή να έχουμε νέες μορφές ε, παραγωγής ενέργειας όπως για παράδειγμα το υδρογόνο για το χάλιβα. Τρίτο παράδειγμα. Η άμυνα. Και εδώ οι νέες τεχνολογίες παίζουν σημαντικό ρόλο. Άλλες περιοχές του κόσμου, άλλα κράτη, επενδύουν ε, τεράστια ποσά για τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της άμυνας. Θέλουμε να συνδυάσουμε τους πόρους μας, να εντοπίσουμε τις κοινέ μας ανάγκες από κοινού, ούτως ώστε και εκεί και στον κλάδο αυτό να διασφαλίσουμε την τεχνολογική κυριαρχία μας και αυτό θα έχει και επιπτώσεις ε, στη μη στρατιωτική βιομηχανία για τι επιχειρήσει και του συμπολίτε, στον ε, πολιτιστικό τομέα. Και εκεί η τεχνολογία παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Δύσκολα μπορούμε να διαχωρίσουμε την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται, φτάνουν στους ε, συμπολίτες μας. Πρέπει λοιπόν να επαγρυπνούμε για να υπάρχει η ελευθερία να ε, ανταποκρινόμεθα στην αντίληψη που έχουμε για τι ε, τις τη Ευρώπη και να προστατεύουμε τη δημοκρατία, του συμπολίτε μα τα παιδιά, ιδιαίτερα προ του Γερμανού συναδέλφου, αλλά και προ άλλου ε, ε, λόγω των θλιβερών γεγονότων του Χάλε. όλοι υποφέρουμε από αυτό που συνέβη. Το μίσο και ο αντισημιτισμό έδειξαν για άλλη μια φορά το φρικαλαίο πρόσωπό του με σύγχρονα μέσα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε και εμεί μέσα τι αναγκαίε απαντήσει απόλυτα ισορροπημένες που μπορούν να μα ε, προσφέρουν οι δημοκρατίε. Επίση, οι νέε τεχνολογίε αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσει, με τον οποίο εργάζονται οι άνθρωποι, πω μαθαίνουν. Δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα στο περιθώριο. Υπάρχει λοιπόν και μια κοινωνική πλευρά. Οπότε είμαι πεπισμένη ότι πρέπει όλα αυτά τα θέματα να τα αντιμετωπίσουμε συνδυασμένα και από κοινού. Γιατί τα θέματα τη τεχνητή νοημοσύνη είναι και θέματα πνευματική ιδιοκτησία. Τα θέματα κυκλικότητα μπορεί να εξαρτώνται και από τι δημόσιε προμήθειε και η διανομή των πολιτιστικών αγαθών σημαίνει κανόνε. Νομίζω ότι οι αρμοδιότητε μου αυτέ μου επιτρέπουν να αποφύγω οποιαδήποτε στεγανά, γιατί πολύ συχνά, στο σώμα αυτό που και εγώ τόσα χρόνια είμαι μέλο, ακούω πολλέ επικρίσεις ότι είναι πολύ γραφειοκρατικέ ορισμένε προσεγγίσεις με διάφορα στεγανά, πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Δύο συγκεκριμένα παραδείγματα, όπου μπορούμε να έχουμε ε, πολύ γόνιμε συνεργασίε. Για τι μικρομεσαίε, για παράδειγμα, μπορούμε να συνδυάσουμε την εργασία των διαφόρων γενικών διευθύνσεων, ούτω ώστε όλοι όσοι ασχολούνται με τι επιχειρήσει, είτε είναι ψηφιακά θέματα, είτε είναι θέματα χρηματοδότηση για τον τομέα άμυνα, είτε είναι θέματα πιο παραδοσιακών πολιτικών, να έχουν ένα συνομιλητή. Επίση, μπορούμε να βοηθήσουμε να συνεργαστούν καλύτερα όσοι ασχολούνται με την εφαρμογή των ε, αποφάσεών μας, ούτως ώστε να μαθαίνουμε ημένα από τους δε, ούτως ώστε η εσωτερική αγορά να αναπτυχθεί περαιτέρω. Επίση, ε, με ρωτήσατε, μα πώ θα διαχειριστείτε τόσο πολλέ αρμοδιότητε. Ε, φυσικά δεν το κάνω μόνη μου, αλλά με την ομάδα μου, με τη στήριξη των υπηρεσιών, με τη στήριξη των συναδέλφων μου, επιτρόπων, με τη στήριξη των αντιπροέδρων, με τους οποίους έχω ειδική εντολή να συνεργάζομαι, εφόσον φυσικά με επικυρώσετε βεβαίως. Κατάλαβα πολύ καλά ότι πρέπει να υπάρχει χρηστή διαχείριση. Ορισμένοι μου είπανε, μα πώς θα τα καταφέρετε, πώς θα διασφαλίσετε ότι οι υπηρεσίες αυτές θα λειτουργούν σωστά, ότι οι δημόσιοι πόροι των ταμείων ε, υπό την αρμοδιότητά μου θα ε, διατεθούν σωστά. Τα άκουσα όλα αυτά, υπενθυμίζω ότι πρέπει να εργαστούμε και έναντι του εξωτερικού κόσμου. Ελπίζω λοιπόν να μου δώσετε την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σας, ξέρω ότι εσείς βοηθάτε να περάσει η γνώμη των συμπολιτών και εγώ επιχείρησα να το κάνω αυτό όταν ήμουν στη θέση σας Οπότε μιλώντας με τους καταναλωτές, τα συνδικάτα, τι επιχειρήσεις, τα εθνικά κοινοβούλια, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ορισμένα θέματα. Ξέρω ότι είναι δύσκολα θέματα, επί των οποίων ορισμένες φορές υπήρξαν ε, συζητήσει ε, πολιτικά φορτισμένες τα τελευταία χρόνια. Μαζί σας λοιπόν θέλω να συνεργαστώ γιατί σε όλη μου τη ζωή ενεθάρρυνα του ε, Ευρωπαίου ε, να συνεργαστούν. Εδώ και 30 χρόνια ασχολούμαι με τι ευρωπαϊκέ υποθέσει. Ε, Πώ περνάει ο χρόνο. Αλλά τα 30 χρόνια ξεκίνησαν τότε με την πτώση του τείχου του Βερολίνου. Τώρα είμαστε σε ένα πλαίσιο ίσω πιο δύσκολο, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει επιτρέψει στην Ευρώπη όλη αυτή η καταπληκτική εξέλιξη, η συμφιλίωση μια ολόκληρη πύρου. Σε όλη μου τη ζωή αυτά τα έκανα, προσπαθούσα να φτιάξω γέφυρε για να συνεργαστούν Ευρωπαίοι. Το έκανα και στο Ινστιτούτο Μπέρ ε, πρέπει να το θίξω γιατί δημιουργήθηκαν πολλά ερωτηματικά στις γραπτές ερωτήσεις σας. Ε, όπως σας είπα, λυπάμαι βαθιά γιατί η δραστηριότητα αυτή των δύο ετών μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολίες για την δέσμευσή μου, για την ακαιρεότητά μου, για την δυνατότητά μου να δρω ανεξάρτητα. Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ε, σε τι βαθμό οι αξίες αυτές είναι για μένα πρότιστες. Και αυτές τις αξίες, αν με επικυρώσετε Αυτές τις αξίες θα προασπίσω με περισσότερη παγρύπνηση, με βάση και την εμπειρία. Όλοι μαθαίνουμε από τις εμπειρίες μας για να προχωρήσουμε. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουμε και το αυστηρό πλαίσιο του κώδικα διοντολογίας. Τώρα το θέμα μιας παρέτησης που αναφέρθηκε. Θα ήθελα να πω τα εξή. Υπάρχει μια πλευρά που είναι σαφώς πολιτική. Είναι μια πολιτική επιλογή που αντιμετωπίζει κανείς όταν ε, έχει ευθύνε. Εάν μου απαγγελθεί κατηγορία που προ το παρόν δεν υπάρχει, μέχρι στιγμή δεν υπάρχει, όπω ή οδήποτε άλλο μέλο του Σώματο των Επιτρόπων, θα συζητήσω με την Πρόεδρο. Γιατί είναι δική τη ευθύνη. Για να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Και από μόνη μου, ή αν μου το ζητήσει, προφανώ, αν είναι αναγκαίο, θα κάνω τα αναγκαία. Αλλά αυτό είναι ο, το δεύτερο στάδιο υπάρχει και μια νομική πλευρά, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και νομομαθείς εδώ. Ε, από πλευράς νομικής, αν δημιουργήσουμε αυτοματισμό μεταξύ της έναρξης μιας διαδικασίας και της ε, παρέτησης, δημιουργείται ένα πρόβλημα. Με δύο πλευρές. Πρώτα απ' όλα πρόβλημα ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπορούμε να την ε, διακυβεύουμε. Διότι υπάρχει ε, οι διαδικασίε στα διάφορα κράτη-μέλη είναι ιδιαίτερα ετερόκλητε. Άρα δεν ξέρουμε σε ποια φάση η ασδήποτε διαδικασία σε κάθε κράτο μέλο θα επελέγεται να παραιτηθεί κάποιο. Άρα δημιουργείται διαφορά αντιμετώπιση των ε, μελών τη Επιτροπή. Και μετά υπάρχει και θέμα τη ε, διαφορά των παραβάσεων. Κοιτάξτε. Θεωρώ ότι πρέπει να καταδικαστεί, πρέπει να παραιτηθεί κανείς όταν καταδικαστεί, αλλά όσο ε, είναι ακόμη κάτι σε ένδικη διαδικασία, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτοματισμός. Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία με ξεπερνούν, αφορούν το σύνολο του Σώματο των Επιτρόπων, το σύνολο των νομικών τάξεων και ε, φυσικά θα συζητήσω με την κυρία Φοντερ Λάιν και με νομομαθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους πολίτες που μας ακούν. Αυτά εισαγωγικά και φυσικά στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Γκουλάρ. Uh, Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ερωτήσεις. Από το ΕΛΚ πρώτα, ο κύριος Κόβατσεφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, κυρία υποψήφια Επίτροπε, θέλω να σας ρωτήσω για το geo-blocking ε, και το σχετικό κανονισμό και τα προβλήματα σχετικά με το πεδίο αυτού του κανονισμού. Ε, είμαστε πολύ κοντά στην προθεσμία τη πρώτη αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντίκτυπο του σχετικού κανονισμού στην εσωτερική αγορά. Και βεβαίω ε, προσπαθούμε να δούμε πώ θα μπορέσουμε αυτοί οι περιορισμοί να μην υπονομεύουν την ενιαία αγορά και τις επιγραμμικές αγορές. Θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση σε αγαθά, σε υπηρεσίες, σε επιγραμμικά στην ε, ε, ψηφιακή αγορά. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε εθνικά σύνορα εδώ. Θα προτείνεται όντω διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής για να συμπεριληφθούν και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρουν περιεχόμενο που προστατεύεται από copyright όπως τα παιχνίδια online, τα βιβλία, τα ηλεκτρονικά, η μουσική κτλ. Ευχαριστώ την κυρία Γκουλά. Η κυρία Γκουλά έχει το λόγο τώρα για να απαντήσει παρακαλώ. Ευχαριστώ ε, για το ερώτημά σας. Νομίζω πως ε, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα της πραγματικότητα αυτή τη ενιαίας αγοράς που γίνεται ψηφιακή αγορά. Όλοι θα δοκιμάσετε να αγοράσετε ένα ε, εισιτήριο αεροπορικό ή να αγοράσετε ένα βιβλίο ηλεκτρονικό και να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα. Ε, πιστεύω ότι η εσωτερική αγορά θα είναι σύγχρονη και ζωντανή μόνο αν βρούμε μια λύση για αυτά τα προβλήματα. Όπως γνωρίζετε υπάρχει ένας κανονισμός που επιτρέπει να μην υπάρχουν διακρίσεις είναι πολύ μικρός ο αριθμός των επιχειρήσεων που όντως αυτή τη στιγμή πολλούν διασυνοριακά ε, επιγραμμικά. Είναι λίγες ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ε, αυτά τα συστήματα. Μου λένε παραγωγή ίνου ότι δεν μπορώ να στείλω ένα κρασί που δοκίμασαν οι τουρίστες το καλοκαίρι εδώ. Μετά από δύο χρόνια είχαμε πει ότι θα γίνει αυτή η αξιολόγηση, οι εργασίες αυτές είναι εξελίξη εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να πάμε προς την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει να εντοπίσουμε τις δυσκολίες. Αναφερθήκατε στο περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Είναι ένα λεπτό ζήτημα, δεν είναι το μόνο. Θα γίνει λοιπόν αυτή η μελέτη σε βάθος και από εκεί και πέρα θα πρέπει να συνεργαστούμε με τις οργανώσεις καταναλωτών, με τον κλάδο, αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να βρεθούν τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μια δεύτερη ερώτηση από τον κύριο Κοβάτσεφ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Μια και μιλάμε για δύο μέτρα και δύο σταθμά στο θέμα αυτό ε, του geo δεν θεωρείτε ότι ε, η κυβέρνησή σας ε, έχει επιλέξει εσάς ε, ως υποψήφια επίτροπο δεν είναι και αυτό δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εσεί είχατε παραιτηθεί ω υπουργό δικαιοσύνη στη Γαλλία. Οι λόγοι για του οποίου παραιτηθήκατε δεν ισχύουν εδώ, στην προκειμένη περίπτωση. κυρία Γκουλάρ. Ναι, να απαντήσω ευχαριστώ. Όπω είπα, πρόκειται για δύο διαφορετικέ ε, περιπτώσει. Εν τω μεταξύ, μετά από δύο χρόνια, ε, η γαλλική δικαιοσύνη με άκουσε, δεν μου είχε απαγγελθεί κατηγορία. Είναι διαφορετική η κατάσταση από νομική πλευρά, από δικαστική πλευρά. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δικό θεσμικό όργανο, αποφάσισε σε μια απόφαση τη Γενική Γραμματεία, μετά από εξέταση σε βάθο ε, τη περίπτωση, ότι ο βοηθό μου είχε εργαστεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε ε, να είναι το θεσμικό όργανο που έχει ζημιωθεί στην προκειμένη περίπτωση. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ είναι πολύ πιο σαφή τα πράγματα. Βεβαίω δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, διότι ο χρόνο τη δικαιοσύνη δεν είναι ο ίδιο με αυτό τη πολιτική ζωή ή τη διοικητική ζωή. Ελπίζω ε, να ολοκληρωθεί γρήγορα αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπορζάν τώρα έχει το λόγο από την ομάδα SD. Ευχαριστώ. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, είσαστε υπεύθυνοι για την πολιτική διαστήματος, για την αμυντική βιομηχανία, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ε, βιομηχανική στρατηγική, εσωτερική αγορά, ψηφιακή, ε, ψηφιακές τηλεπικοινωνίε, ε, ΜΜΕ, οπτικοακουστική πολιτική. Στι σημερινέ σα απαντήσει και στον λόγο σα, είπατε ότι θέλετε να αυξήσετε τι συνεργασίε ανάμεσα στι τρει γενικέ διευθύνσει και να βασίσετε τι πολιτικέ σα και τι προτάσει σα στον τομέα των, ε, του οπτικοακουστικών, των ΜΜΕ, των ε, υπηρεσιών κτλ. σε διαβούλευση. Και μόνο, μόνο και μόνο το να διαβουλευτείτε με όλους αυτούς χρειάζεται χρόνος. Μόνο και μόνο για να επισκεφτείτε τις πρωτεύουσες των κρατών μελών και να έρθετε σε επαφή με το Κοινοβούλιο και να διαβουλευτείτε με τις διάφορες εμπλεκόμενες επιτροπές, χρειάζεται χρόνος. Όλο αυτό το άχθος εργασίας, πώς θα το βολέψετε, και πώς ε, όλες αυτές τις απόψεις θα τις κάνετε συγκεκριμένες δράσεις και θα δώσετε αυτά αποτελέσματα για την Ευρώπη. Πώς θα αντιμετωπίσετε με ισότιμα τα τρία χαρτοφυλάκια, θα δώσετε την ίδια προσοχή στους διαφορετικούς τομείς, δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι, οποίοι πιέζουν και επίγουν. Κύριε Γκουλάγ, ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Κοιτάξτε, ξέρω ότι πρέπει να δουλέψω και δεν είμαι η μόνη. Όταν ήμουν στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και είχα απέναντί μου επιτρόπους που είχαν την ευθύνη του ευρώ, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της φορολογίας, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολλά να κάνουν. Ε, δεν φοβάμαι να αναλάβω ένα τόσο βαρύ χαρτοφυλάκιο. Όταν επισκεπτόμαστε τις πρωτεύουσε, επισκεπτόμαστε τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, των συνδικάτων, κάλλιστα, ε, εκπροσώπους στο ΜΜΕ, στα Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να υπάρχουν βουλευτές που ασχολούνται με διαφορετικά θέματα. Το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Αν προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε γέφυρες και δεσμούς, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, να καλύψουμε πολλά θέματα. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική προσέγγιση. Αυτό προσπάθησα να σας πω στην εισαγωγή μου πρέπει να κοιτάξω κάποια θέματα από τη σκοπιά του, του ψηφιακού τομέα, γιατί αυτή είναι και η ευθύνη μου. Θα είδατε και την ε, διοργάνωση και την οργάνωση του Σώματος του Επιτρόπου για τα ψηφιακά. Η Μάργαρετ Βεστάγκερ, η Αντιπρόεδρος, θα παίξει ρόλο. Ο Βάλης Ντομπρόσκη είναι επιφορτισμένος με θέματα με τα οποία θα ασχοληθώ και εγώ, είναι άτομα που γνωρίζω. Ειδικά όταν ασχολιόμουν με τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα και τα ήξερα όταν δούλευα στη Τράπεζα τη Γαλλία. Του ήξερα. Θα έχουμε μια ομάδα που θα συνεργάζεται. Όσο περισσότερο μπορεί. Δεν είναι απλό. Έχετε δίκιο. Θα ήταν αλαζονικό να πω ότι είναι εύκολο να τα καταφέρω. Να σας πω και κάτι πιο προσωπικό είναι όπως όταν έχουμε πολλά παιδιά. Εγώ έχω τρία παιδιά. Πάντα προσπάθησα να δώσω και στα τρία απεριόριστο χρόνο. Μερικές φορές είναι εύκολο, μερικές φορές είναι πιο δύσκολο. Κάποια στιγμή κάποιο χρειάζεται περισσότερη φροντίδα. Θα προσπαθήσω να κάνω το ίδιο και ελπίζω να ότι θα με στηρίξετε. Ευχαριστώ πολύ. Ασυμπληρωματική ερώτηση, κύριε Μποζάν. Ένα μικρό σχόλιο. Ελπίζω προ όφελο των Ευρωπαίων, εάν περάσετε αυτή την ακρόαση, να μην χρειαστεί να σας πούμε «εμείς σας τα λέγαμε». Τώρα για τη συμπληρωματική ερώτηση. Έχετε ένα βασικό στόχο να μειώσετε την, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να φτάσετε σε μηδενικές εκπομπές. Ε, αλλά για το θέμα αυτό έχουμε άλλον επίτροπο και πολύ σωστά έχουμε διαφορετικό επίτροπο. Οι πολιτικές είναι αλληλένδετες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τα αναλάβει όλα ένας επίτροπος. Αυτό θα πρέπει να το πετύχουμε μέσω συντονισμού και συνεργασίας, αντί μέσω της διαβούλευσης που μπορεί να υποσκάψει τον ηγετικό ρόλο, τον έλεγχο και τη γνώση του χαρτοφυλακίου. Αυτές οι τεράστιες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε δεν νομίζω ότι χρειάζονται προσοχής, της προσοχής πάνω από ένα ατόμου δεν υπάρχει κίνδυνος να μην δώσετε αρκετή προσοχή ε, σε τομείς του χαρτοφυλακίου σας, όπως παραδείγματος χάρη στα ΜΜΕ και στον πολιτισμό. Το πρόγραμμα Media, ας πούμε, για ποιο λόγο να είναι στο ίδιο χαρτοφυλάκιο με τα προγράμματα της άμυνας. Η κυρία Γκουλάχ. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Το είπατε κι εσείς. Είναι ευρύ το χαρτοφυλάκιό μου, αλλά δεν καλύπτει και τα πάντα. Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής αυτής είναι να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα και η ευρωπαϊκή οικονομία τουλάχιστον να ακολουθήσει αυτή την τραπώ. Ε, ο Τίμερ μας θα ασχοληθεί με αυτό ε, και ο Επίτροπος που θα ασχοληθεί με το περιβάλλον και τους ωκεανούς είναι υπεύθυνοι για αυτά. Αυτή τη συνεργασία, αν δείτε το πώς είμαστε οργανωμένοι, θα την προωθήσουμε. Ο κάθε Επίτροπος παρεμβαίνει σε θέματα του άλλου, γιατί με αυτόν τον τρόπο απεικονίζεται και η διαφορετικότητα των απόψεων και των πολιτισμών. Έτσι εκπροσωπούμε τις πολιτικές μας οικογένειες και τις χώρες μας. Για τα ΜΜΕ και τον πολιτισμό. Δεν έφτιαξα εγώ το χαρτοφυλάκιό μου, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε εκ των προτέρων να πω ότι θα ασχοληθώ μόνο με το α θέμα και όχι με το β. Αν υπάρχουν προσαρμογέ που πρέπει να γίνουν, φυσικά θα πρέπει να τι κάνει η κυρία Φόντερ Λάιεν. Εγώ δεν έχω την πρόθεση να παραβλέψω τον πολιτισμό. Το είπα και την προηγούμενη φορά. Πιστεύω ότι ο πολιτισμός είναι μέσω χειραφέτησης των ατόμων. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να φέρουμε σε αντιπαράθεση τα θέματα άμυνας, πολιτισμού και βιομηχανίας. Θα πρέπει να διαχειριστούμε όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα, τις ανάγκες της κοινωνίας που θέλει και να προστατευτεί από τις εξωτερικές επιθέσεις, αλλά και που θέλει να προστατεύσει τα στοιχεία ταυτότητά τη, που είναι ο πολιτισμό τη και η γλώσσα τη. Δεν νομίζω ότι το ένα έρχεται σε αντίθεση με το άλλο. Το ένα αποκλείει το άλλο. Ζωβά. Στο κυρία Σαραντζοβά από το Ρινιού. Ευχαριστώ. Αγαπητή Σιλβή, οι συνάδελφοι ήθελαν να υπάρξει μια δεύτερη ακρόαση για να ακούσουν ε, καλύτερα τις ιδέες σας για την ενιαία ώρα. Ελπίζω ότι αυτή η ακρόαση θα σας το επιτρέψει λοιπόν αυτό. Κανείς δεν αφισβητεί την ισχυρή δέσμευσή σας ε, για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και είμαι πεπισμένη ότι έχετε και με το παραπάνω τα απαραίτητα προσόντα για να γίνετε επίτροπος. Έχετε όλα τα προσόντα για το χαρτοφυλάκιό σας. Τώρα, δεν πρέπει να είναι κανείς αφελής όσον αφορά τα εμπορικά συμφέροντα και τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών. Από ό,τι καταλαβαίνω, σε διάφορα κράτη-μέλη η κοινή γνώμη θέλει να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Αλλά θα ήθελα να μάθω εάν θεωρείτε ότι η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα θέσει σε ε, ε, μειονεκτική θέση τη επιχειρήση μα έναντι των Αμερικανικών και Κινέζικων. Ποια είναι η άποψή σα, πώ μπορείτε να με καθησυχάσετε. Είναι σημαντική η ερώτησή σας. Χαίρομαι που θέτετε το θέμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει μετάφραση στα γερμανικά. Λοιπόν, Ναι, μπορώ να τα πω γερμανικά, αλλά δεν τα καταλαβαίνουν οι άλλοι, λέει η κυρία Κουλά. Αν μίλαγα αγγλικά συνέχεια, θα μου λέγατε ότι δεν ασχολούμαι με την κουλτούρα. Η κουλτούρα είναι επίση η πολυμορφία. Αυτό που θέλω να πω στην κυρία Σαράντζοβα είναι το εξή. Ευχαριστώ που θέσατε το θέμα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει πρόβλημα με τα γερμανικά.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 I hope it was functioning until now. Ελπίζω να λειτουργούσε νωρίτερα. No, no. Okay ναι, παρακαλώ, κυρία Γκουλάρ, μπορείτε να αρχίσετε και πάρετε την απάντησή σα. Ναι, για όσου το άκουσαν, συγγνώμη που τα επαναλαμβάνω. Ήθελα να πω λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό στη συζήτηση αυτή να μπει αυτή η παγκόσμια, η σφαιρική αντίληψη. Βρισκόμαστε σε μια καμπή και γι' αυτό αναφέρθηκα στην τεχνολογική ανατομία αρχικά. Βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή όπου οι καινούριε επιχειρήσει μα, οι startup, είναι πάνω από 10.000 που ασχολούνται με το ψηφιακό τομέα και που έχουν ανταγωνιστούν με γίγαντες, με εταιρείε που ενδεχομένως να μπορούν να καταχραστούν της εξουσία τους, που έχουν έναν αριθμό δεδομένων πολύ σημαντικό και αυτές οι εταιρείε είναι κατά μεγάλη πλειοψηφία αμερικανικές και κινέζικες για την ώρα. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ λοιπόν, εφόσον με εμπιστευτείτε, με την, υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να ξεχρονίσω το νομικό πλαίσιο που αυτή τη στιγμή είναι κατακαιρματισμένο, που δεν είναι ασφαλές και που δεν είναι προσαρμοσμένο απέναντι στην πρόκληση αυτή. Βεβαίως υπάρχουν ζητήματα ανταγωνισμού, ε, θα πρέπει να δούμε πώς αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις έρχονται εδώ, αλλά θα πρέπει πάνω απ' όλα να σεβαστούμε τις αρχές μας, την αρχή της χώρας προέλευσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε στο ιστορικό της ενιαίας αγοράς να εξυπηρετούμε το σύνολο της αγοράς ε, βρισκόμενη σε μία χώρα. Υπάρχει επίσης η αρχή της ευθύνης των πλατφόρμων αυτών και η αρχή της ελευθερίας έκφρασης επιγραμμικά. Βεβαίως, από την άλλη, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κατακρεματισμό. Πολλά κράτη-μέλη ε, έχουν εγκρίνει νομοθετήματα τα οποία αποκλίνουν μεταξύ τους. Θα πρέπει επίσης να μπορούμε να εντοπίσουμε ε, το παράνομο ε, περιεχόμενο. Δεν θέλω να εκμεταλλευτώ αυτό που συνέβη χθε βέβαια γιατί δεν θα ήταν σωστό. Αλλά είναι άλλο ένα παράδειγμα ε, της χρήσης της επιγραμμικής περιεχομένου μίσους και πράξεων μίσους. Θα πρέπει να βρεθεί λοιπόν το σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ της ελευθερίας που επιθυμούμε τη διευκόλυνση του συνοριακού εμπορίου, της δυνατότητας ανάπτυξης του ψηφιακού αυτού τομέα και από την άλλη ε, να προστατεύσουμε αυτό που πρέπει να προστατευτούν. εγώ δεν θέλω επιγραμμικό έλεγχο ή έλεγχο της σκέψης, αλλά θα πρέπει να ελέγχουμε όσους από μόνοι τους ε, δρούν παράνομα και επίσης ε, έχουν ένα λόγο μίσους και προωθούν τη βία. Η κυρία Σαράζο θέλει να επανέλθει με κάποιο δεύτερο ερώτημα. Ναι, σα ευχαριστώ πολύ για τη σαφέστατη απάντησή σας. Θα ήθελα να αναπτύξω λόγο περισσότερο το ερώτημά μου. Αναφερθήκατε στον κατακαιρματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς ε, σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό τομέα. αλλά και την νομοθεσία και το πώς αυτή επηρεάζει τους μικρούς παίχτες. Πώς λοιπόν αυτή η ψηφιακή αγορά δεν θα πλήξει αυτούς ε, τους μικρούς παίκτες, τις μικρές επιχειρήσεις. Η κυρία Ναι, ακούστε, εδώ πάλι δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια, αλλά είναι σημαντικό να επιμείνω. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια συνοχή στη δράση μας. Μια μικρή επιχείρηση είναι μια μικρή επιχείρηση, είτε δρά ψηφιακά, ε, στον ψηφιακό κόσμο, είτε όχι. Τα χρήματα λοιπόν, τα μέσα που διαθέτουμε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εδώ. Το να έχουμε ένα προπολογισμό ε, που θα ε, βοηθάει τι επιχειρήσει αυτέ, να υπάρχει ένα εκπρόσωπο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ε, είναι καλέ ιδέε. Στον ψηφιακό τομέα αυτό μπορεί να μα οδηγήσει στο να πάρουμε μια σειρά από αποφάσει ρυθμιστικού τύπου, διότι θέλουμε να ξεχρονίσουμε το ευρύτερο πλαίσιο, αλλά και εφαρμοστικού διότι ενδεχομένω κάποιε χώρε μπορεί να μην μεταφέρουν σωστά κάποια νομοθετήματα, κάποιε νομοθετικές πράξει ή που δεν θα φροντίσουν οι μικρέ επιχειρήσει να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον τομέα και να δραστηριοποιηθούν εκεί. Πρέπει να συνδυάσουμε λοιπόν τα διάφορα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα ρύθμιση, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και υπάρχει βεβαίω προβλέπονται ειδικά, ειδικά κονδύλια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το επίπεδο τη εφαρμογή, βέβαια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Κάεμ από τους Πράσινους. Κύριε Γκουλάρ, πέρα από τις διαφωνίες μας επί της ουσίας, ε, η ομάδα μου έχει δύο μεγάλες ανησυχίες για την ε, ηθική και, τις δια... και τη διάσταση του χαρτοφυλακίου από την ε, εσωτερική αγορά μέχρι την άμυνα. Έχουμε επιφυλάξει παρά τις διευκρινήσεις. Αλλά η υποψηφιότητά σας είναι πραγματικά πρόβλημα δεοντολογίας. Και επειδή είμαστε στο Brexit δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και του εκπροσώπου ή τι εκπροσώπου. Οι γραπτέ σα απαντήσει και οι εξηγήσεις σήμερα το πρωί δεν μα καθησύχασαν. Λυπάστε, είπατε, ότι η δραστηριότητα που είχατε παράλληλα ε, με την δραστηριότητα βουλευτού δημιουργεί αμφιβολίε. Καταλαβαίνετε και δέχεστε ότι δεν είναι δυνατόν ε, ένας όμιλος ε, προβληματισμού να σα πληρώνει όσο σα πληρώνει και το δημόσιο. Το πρόβλημα ηθικής δεν το διαπιστώσατε παρά μόνο αναδρομικά. Πώς θεωρείτε λοιπόν πως έχετε την αναγκαία ακαιρεότητα για να ασκήσετε τα καθήκοντά σας. Μήπω θα έρθετε σε πέντε χρόνια να μα πείτε ότι και πάλι αναδρομικά θα έπρεπε να τα έχετε κάνει κάπω διαφορετικά τα πράγματα. Ευχαριστώ, κύριε Αγκούλα. Κύριε συνάδελφε, αυτό που προσπάθησα να απαντήσω με τις ερωτήσεις μου είναι ότι από τη μία μεριά υπάρχουν κανόνες δικαίου και από την άλλη μεριά υπάρχουν θέματα διοντολογίας και δίκης. Σέβομαι βαθιά αυτά που είπατε για τα θέματα της διοντολογίας. Είχα την ευκαιρία να το συζητήσω με διάφορα άλλα μέλη της ε, πολιτικής σας και το συζητώ και σήμερα μαζί σας. Ε, αυτή η διαφορά είναι ότι το δίκαιο επιτρέπει ορισμένα πράγματα και τα επιτρέπει ακόμη, επέτρεπε και το επιτρέπει, οι βουλευτές να έχουν κάποια άλλη δραστηριότητα. Είναι μια, ένας όμιλος μελετών, ιδιωτικός, αλλά ο οποίος ε, προωθούσε ιδέες υπέρ της Ευρώπης και τα άτομα με τα οποία συνεργαζόμουν είναι άτομα τα οποία εκφράζονται σαφώς υπέρ της Ευρώπης. Η ηθική, η είναι ένα θέμα κάπως ε, πιο υποκειμενικό. Τα διάφορα άτομα αντιλαμβάνονται αυτά τα θέματα διαφορετικά. Άρα είναι πολύ λεπτό το θέμα όταν ε, έχουμε φύγει από το τομέα του δικαίου. Γιατί εκεί υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, όπως είπα στην απάντησή μου. Αυτές οι ερωτήσει, πρέπει πάντα να τίθενται. Τώρα βεβαίω υπάρχουν υψηλότερε απαιτήσει. Ε, θυμάμαι τι μάχε που έδωσε το Κοινοβούλιο για τον κώδικα διοντολογία, για την πρόσβαση των ε, εκπροσώπων ομάδων πίεση, των λόμπι. Αυτά τα θέματα εξελίσσονται. Δεν είναι τίποτα απόλυτα καθορισμένο μια για πάντα. Τώρα πια που ήρθε η στιγμή να διευκρινίσω την κατάσταση. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει ένα σαφή κώδικα διοντολογία. Οι Επίτροπη πρέπει να είναι απόλυτα ανεξάρτητοι και από την πλευρά μου δεσμεύομαι ενώπιον σας να είμαι. Και τώρα, σε ανθρώπινο επίπεδο. Νομίζω ότι όλοι αντιμετωπίζουμε παρόμοιες καταστάσεις, όλοι μπορούμε να μάθουμε από τις εμπειρίες μας. Ελπίζω ότι και εγώ θα μάθω και θα αντιμετωπίζω τις καταστάσεις ε, με περισσότερη πείρα βεβαίω, ε, Οι άνθρωποι κάνουν τις ιδέες και δικαίου και οδοντολογίας να εξελιχθούν. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε και εμένα να εξελιχθώ εγκρίνοντάς με σήμερα. Ευχαριστώ στην πραγματική ερώτηση, κύριε Καρέμ. Ε, ένας άλλος ε, τομέας αφιβολίας. Καταλαβαίνω. Λέτε ότι είστε υπέρ της Ευρώπης. Αλλά λέτε ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές ε, προδιαγραφές αν είναι κανείς ε, πολιτικός σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο ε, Γαλλίας. Γιατί Παρετηθήκατε όταν προέκυψε το θέμα αυτών των αργομιστιών του Μοντέμ, ενώ σήμερα προτείνεται να γίνετε επίτροπος, ε, ενώ υπάρχει διαδικασία να εξελίξει. Βεβαίω δεν σα έχει απαγγελθεί κατηγορία, αλλά υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο ότι διεξάγεται έρευνα. Απαντήσατε στην πρώτη ακρόαση ότι η διαφορά έχει να κάνει με το ότι το γεγονό ότι δεσμεύεστε είναι σοβαρότερο. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δεν θα έπρεπε να παραιτηθείτε εάν σα απαγγελθεί κατηγορία, ενώ θα το κάνατε αν είσαστε υπουργό στη Γαλλία. Η κυρία Γκουλά. Καταρχάς, συγγνώμη που θα χρειαστεί να επαναλάβω αυτό που επιχείρησα να εξηγήσω απαντώντας άλλη ερώτηση. Υπάρχουν δύο θεμελιώδεις διαφορές σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017. Πρώτα απ' όλα, ο Γενικός Γραμματέας αυτού του θεσμικού οργάνου έκανε διοικητικούς ελέγχους και κατέληξε ότι ο βοηθός μου είχε εργαστεί για πάνω από πέντε χρόνια και υπήρξε μια δυσχέρεια που είχε να κάνει με τον τρόπο παρέτησής του γιατί συμφωνήσαμε μια, ένα φιλικό διακανονισμό αντί μιας διαδικασίας πιο βαριάς και πιο δυσάρεστης. Οπότε νομίζω ότι αυτό με καθησυχάζει. Είστε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, μπορείτε να ρωτήσετε τον Γενικό Γραμματέα σας που θα βεβαιώσει, όπως είπε και δημοσίως στον τύπο, ότι το θέμα έχει λήξει. Βεβαίως έχετε δίκιο, δεν έχει εκφραστεί ακόμη δικαιοσύνη. Και γι' αυτό είμαι ακόμη επιφυλακτική, αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο προέκυψε από το ίδιο το θεσμικό οργάνο που θα μπορούσε να πει «Μα έχουν θυγεί τα συμφέροντά μου». Επίσης, τον περασμένο Σεπτέμβριο, δηλαδή πάνω από δύο χρόνια, γιατί έτσι προχωράνε οι δικαστικές ε, έρευνες κατέθεσα εθελουσίω και δεν υπήρξε καμία αλλαγή στο καθεστώ μου. Βεβαίω, έχετε δίκιο, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα μετρημένη. Αλλά φυσιολογικά δεν νομίζω ότι θα μου απαγγελθεί η κατηγορία. Αυτά νομίζω ότι είναι κάποια στοιχεία και με συγχωρείτε, αλλά ήδη ξεπέρασα αρκετά τον χρόνο. Ευχαριστώ η κυρία Ζωγόν τώρα από την ΙΝΤΕ. Ναι, είπατε ότι είστε καθαροί ε, και το 2013 είχατε πει ότι δεν έχει σημασία, δεν, έχετε, δεν είχατε κάποιο σημαντικό ρόλο. 13 εκατομμύρια ε, το μήνα βγάζει αυτή η εταιρεία στην οποία εργαστήκα το σύμβουλος. Ε, διαβάζω εδώ τις νέες απαντήσεις σας, πάλι για την ακαιρεότητα δεν μας τα λέτε καθαρά. Οι αποφάσεις σας είναι αμφίσιμες, οι απαντήσεις σας είναι αμφίσιμες. Γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ και σας θέτουμε ξανά ερωτήματα μας. Είπατε ότι δεν ήσασταν ε, εργαζόμενοι μισθωτοί σε αυτό το λόμπι, όμως είχατε μια ε, σύμβαση συμβούλου από αυτό, με αυτό το think tank και αναφερθήκατε στο Ινστιτούτο Μπεργκρούεν. κυρία αντι, του, της τραπέζας της Γαλλίας, πού είναι η αποστολή που είχατε αναλάβει, πού ε, είναι ε, ο μισθό σα, ποιο είναι το νομικό καθεστώ τελικά βάσει του οποίου πληρωθήκατε από αυτό το think tank. Και η κυρία Γκουλάρ, ακούστε κυρία μου, θα επαναλάβω για άλλη μια φορά μια σειρά από πράγματα. Να, φυσιολογικό είναι αυτό. Ε, Αυτή είναι η κανόνε του παιχνιδιού. Δικαίωμά σα είναι να θέτετε τα ερωτήματα. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε μια κατάσταση μισθωτού στη Γαλλία αυτό σημαίνει ότι κάποιος ε, υπόκειται σε έναν ε, εργοδότη και μια, ένα άλλο καθεστώς, αυτό του συμβούλου, όπου περιστασιακά συνδράμω για κάποια ζητήματα. Δεν πρόκειται λοιπόν ε, για εταιρεία, πρόκειται για ένα think tank που οργανώνει ε, συναντήσεις με τους πολίτες για την προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας. Στην απάντησή μου έχω δώσει κάποια στοιχεία συγκεκριμένα. Ε, τα έχουν ε, επιβεβαιώσει αυτά οι άνθρωποι με τους οποίους εργάστηκα. Νομίζω ό,τι είχα να παρουσιάσω το θέμα αυτό, τα παρουσίασα. Κατά τα λοιπά, ε, σας παραπέμπω στις γραπτές μου απαντήσεις. Ναι, ευχαριστώ. Μια δεύτερη ερώτηση. Κυρία Ζωγόν, παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά τα δραστηριότητά σα, αυτό το think tank, ε, στι γραπτέ σα απαντήσει, τι να πω. Πώ ήταν σε επαφή, ετοιμάζατε τα τηλεφωνήματα, την σα διάταξη, του ε, συμμετέχοντε και λέτε ότι από το δεύτερο εξάμεινο του 2015 συνεργαστήκατε με τον Κίφερ Χόφστατ για να μπορεί αυτό το Συμβούλιο για το Μέλλον της Ευρώπης ε, να μπορέσει ε, να επηρεάσει την, ε, το, το δημοψήφισμα για τον Brexit, όταν είχε ακόμα ανακοινωθεί τότε το δημοψήφισμα για τον Brexit του κυρίου Κάμερον. Δηλαδή, ουσιαστικά έχετε πληρωθεί για να συνεργαστείτε με τον κύριο Βερχόφστατ, που είναι επικεφαλή ε, τη πολιτική σα ομάδα. Και αυτό είχε κάποια έσοδα από αυτή τη συνεργασία. Τελικά, πώ έλαβε χώρα αυτή η συνεργασία με το Think Tank. Ο Πίτερ Σάδερλαντ ε, και πρόεδρο τη Πολυεθνική Goldman Sachs, τι ρόλο παίζει σε αυτή τη διαδικασία. Κυρία Γκουλάρ, παρακαλώ. Ακούστε, για το δημοψήφισμα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω το 2015 στο πρόγραμμα του Συντηρητικού Κόμματος είχε προβλεφθεί το δημοψήφισμα ως ε, πρόταση. Δεν ήταν λοιπόν επιστημονική φαντασία. Ήδη το Φεβρουάριο του 2016 υπήρχε, υπήρχε συμφωνία μεταξύ η Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Ηνωμένου Βασιλείου για να παρεμποδιστεί αυτό το δημοψήφισμα. Ε, να υπάρξει μια νέα νομική βάση, εν πάση περιπτώσει, ε, για τις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν λοιπόν το θέμα αυτό το 2015 ήδη εξαιρετικά επίκαιρο και, και εξαιρετικά σημαντικό. Μιας και εδώ μιλάμε για την παρουσία ενός κράτους μέλους εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια μεγάλη δημοκρατία, ένας μεγάλος σύμμαχος ένας ε, οικονομικός εταίρος εξαιρετικά σημαντικός και ήταν εντελώς φυσιολογικό να ασχοληθώ με το ζήτημα αυτό ε, και δεν το μετανιώνω. Πολλά κόμματα, κινήματα προσπαθούν να επηρεάσουν την απόφαση προς την άλλη κατεύθυνση. Είναι σημαντικό λοιπόν και οι φιλοευρωπαίοι να κάνουν από τη μεριά τους ό,τι μπορούν. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Κράσνοντεύσκη από το ECR. Ευχαριστώ. Προβλέπετε να έχετε πολλές αρμοδιότητες. Άρα και πολλά ερωτήματα θα μπορούσα να θέσω. Ωστόσο, να σας ρωτήσω με κάτι, για κάτι σχετίζεται με το ότι έχετε δημοσίευσει πολλά βιβλία, έχετε ασχοληθεί με τις πολιτικές επιστήμες. Ποιο μοντέλο κοινωνίας και δημοκρατίας θέλετε στην Ευρώπη. Πιστεύετε ότι ένα σύστημα όπου πλούσιοι οι οποίοι ασχολούνται με συζητήσιμες δραστηριότητες μπορούν να επενδύσουν πάρα πολλά χρήματα σε προεκλογικές εκστρατείες για να διαμορφώσουν ε, τη συνείδηση της κοινή γνώμης. Είναι αυτό καλό μοντέλο για την Ευρώπη. Δεν σας ανησυχεί ότι υπάρχουν πολλά επίπεδα επιρροή στην κοινωνία. Δεν θεωρείτε ότι τέτοιες πρακτικές δεν θα πρέπει να ε, αποτελούν τμήμα του μοντέλου μας. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά, λέτε τι οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο εγκρίνω. Εγώ συμφωνώ με το οικονομικό μοντέλο που περιέχεται στις συνθήκες και στο χάρτη, στη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων, δηλαδή η κοινωνική οικονομία της αγοράς. Υπάρχουν αξίες τις οποίες προσυπογράφουν όλα τα κράτη-μέλη που εντάσσονται στην Ένωση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν πρόκειται κάθε φορά να επαναπροσδιορίζουμε τις αρχές μας. Και για μια επίτροπο, αυτά τα δύο κείμενα, οι συνθήκες και η χάρτα θεμελιδών δικαιωμάτων, είναι ο μπουσουλάς μου. Και το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας είναι η παραπληροφόρηση, αν κατάλαβα καλά, η χρήση των νέων μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας, ούτω ώστε κάποιοι ξένοι να επηρεάζουν τη δημόσια ζωή της Ένωσης. Επί του θέματος αυτού έχει ήδη ασχοληθεί η απερχόμενη επιτροπή. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνα, ε, έκαναν μια εξέταση του θέματος αυτού. Είναι πολύ σημαντικό όσοι επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν τις δημοκρατίες μας από απ' έξω, να μην ε, επιτυχάνουν. Αυτά όμως θα τα δω με την κυρία Ζιούροβα και με άλλους αντιπροέδρους και επιτρόπους, γιατί το θέμα αυτό είναι οριζόντιο. Θίγει πολλούς τομείς και απόλυτα θεμελιώδες. Και να μην γελιόμαστε. Μπορούμε να εντοπίσουμε τις δυνατότητες εξωτερικής παρέμβασης και να καταγγείλουμε τα ψεύτικα νέα, την παραπληροφόρηση, τη συκοφάντηση, την αποσταθεροποίηση ούτω ώστε όλα αυτά να μην θίξουν την ανεξαρτησία τη Επιτροπή. Αν κατάλαβα καλά, επαναλαμβάνω την ερώτησή σα. Κύριε Κρασνοντεύσκη, συμπροματική. Κοιτάξτε. Δεν πρόκειτο για κάποιους πολιτικούς, αλλά άτομα με μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, πλούσιοι, οι οποίοι υποτίθεται πω ε, κάνουν φιλανθρωπικέ δράσει, ενώ στην πράξη θέλουν να επηρεάσουν τι πολιτικέ μα διαδικασίε. Δεν θεωρείτε ότι συμπεριφορά ορισμένων ελίτ και υπάρχουν και αμφιβολίε για το δικό σα θέμα, που, για, για εσάς που έχουν να κάνουν με εσά. Δεν θεωρείτε ότι ορισμένα μέλη των ελίτ έχουν μία δράση που είναι στην ουσία κάτι σαν τον λαϊκισμό. Υπάρχει αυτή η κρυφή εξουσία που κρύβεται πίσω από τα think tank, και διάφορες παρόμοιες. Ε, πρόσωψη, φιλανθρωπική, στην πράξη προσπάθεια επηρεασμού της πολιτικής μας διαδικασίας. Η κυρία Γουλά. Α, κατάλαβα καλύτερα τώρα. Κοιτάξτε, σε ένα κράτο δικαίου το μόνο που μετράει είναι ο σεβασμός του νόμου. Από όλους. Οι κοινωνίες μας είναι άνοιχτες, φιλελεύθερες, δεν είναι λοιπόν από μόνο του καταδικαστέο να θέλει να προωθήσει κανείς ιδέες, να ε, συσπηρώνονται και να δρουν από κοινού όσοι θέλουν να το κάνουν αυτό. Αν η συμπεριφορά αυτή μετατραπεί σε παρέμβαση στη δημοκρατία, σε απόπειρα αποσταθεροποίηση, τότε βέβαια αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά εγώ πιστεύω απόλυτα στη δημοκρατία. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι όσοι έχουν ε, φιλανθρωπική δραστηριότητα θα πρέπει να καταδικάζονται. Και μάλιστα συλλήβδην. Νομίζω ότι ό,τι είναι παραπληροφόρηση, ό,τι είναι διάδοση ψευδών ειδήσεων, ό,τι είναι προσπάθεια περιερασμού της κοινή γνώμης, πρέπει φυσικά να καταδιωχθεί χωρίς ε, δισταγμούς. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μπομπάχ, από την το 2017 σε μία συνέντευξη στο Φιγκαρό είπατε ότι θέλετε να αποκαταστήσετε την εμπιστοσύνη και να δώσετε ε, στους ανθρώπους ε, νέα διάθεση για να πιστέψουν στην Ευρώπη. Ε, μπορείτε να συνεισφέρετε. Σκεφτείτε αυτοί, αυτούς που πάσχουν από την ε, λιτότητα. Εσείς ως Επίτροπος θα μπορούσατε να τους αποκαταστήσετε αυτή την εμπιστοσύνη όταν παίρνετε 12.000 ευρώ ε, για να προωθήσετε κάποιους σκοπούς. Ε, πιστεύετε ότι όταν έχετε πάρει 330.000 ευρώ από, τον, από κάποιον πλούσιο, ε, φανταστείτε αυτούς που καταγγέλνουν τα λόμπι στην Ευρώπη. Ε, όταν έχουμε μια πρώην ε, ευρωβουλευτήνα η οποία ε, στην πραγματικότητα προωθούσε ιδέες των λόμπι, μπορούν να την εμπιστευτούν. Επίσης, έχετε σχέσεις με το Ινστιτούτο Μπεργκρούεν. δεν θα έπρεπε σήμερα, μόνο και μόνο αν ήσασταν υπεύθυνοι, να παραιτηθείτε από την υποψηφιότητά σας, κύριε Αγκουλά. Μπορούμε να παρουσιάσουμε τα πράγματα και έτσι και αλλιώ. Μπορούμε κάλλιστα να ρίξουμε λάσπη σε κάποιον ο οποίο πολέμησε για κάτι σε όλη του τη ζωή και να σκεφτούμε ότι απλώς ε, είχε ένα συμβόλαιο δύο χρόνων από... με κάποιον. Επί πολλά χρόνια ε, ήμουνα εδώ στο Κοινοβούλιο και έκανα προσπάθεια για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια ε, στην Καριτάς, σε πολλές άλλες οργανώσεις δούλεψα για να καταπολεμήσω τη φτώχεια η Σίλβια Κώστα, η κυρία Φοντανιέ και άλλοι παλιοί ευρωβουλευτέ μπορούν να το μαρτυρήσουν αυτό. Η Τζίνα Λάμπερτ από του Πράσινου, που ήταν πολύ δραστήρια από το Ηνωμένο Βασίλειο, επίση συνεργάστηκε μαζί μου. Ε, και πάντα θεωρούσα ήταν σημαντικό να ακούσω του ενδεεί, του ε, ξεχασμένου, να του δώσω φωνή σε αυτό το κοινοβούλιο. και ο τον Ντομπρόφσκης και ο κ. Κορές κάνανε τέτοιες προσπάθειες, συνεργάστηκαν μαζί μου. Ε, συνεργάστηκα με ερευνητέ που έχουν γράψει και βιβλία που δείχνουν ότι η πολιτική καταπολέμηση της φτώχειας ε, είναι πολύ καλύτερη όταν ε, την φτιάχνουμε σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους. Είμαι εδώ ενώπιόν σας και σας ζητώ να λάβετε υπόψη όλη μου τη διαδρομή, όλη μου τη σταδιαδρομή. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να μην σας αρέσουν και κάποια που σας αρέσουν περισσότερο. Αλλά αυτή είναι η ζωή μου. Πάντα πολέμησα. Σε κάποιο tweet νομίζω ότι είπατε ότι θα μπορούσαμε να συνοηθούμε τελικά για την Ευρώπη. Σας μιλάω σοβαρά. Αυτό που ήθελα επί πολλά χρόνια σε αυτή την ομάδα, τη διαπραταξή ομάδα κατά πολέμηση της φτώχειας, ήταν να δουλέψω με όλες τις ομάδες. Ε, και με ανθρώπους από την ΚΟΕ. Και στα πλαίσια της ΕΚΟΝ επίσης προσπαθήσαμε να προωθήσουμε τους, τα, τα συμφέροντα των πλέον ενδεών και ελπίζω όλη αυτή η προσπάθεια να μην θεώρησε ότι ήταν ανώφελη. Δεν την καταλάβα την ερώτησή μου. Εγώ δεν επιτίθεμαι στις πεπιθήσεις σας ή στην προσωπική σας ταδιοδρομία. Το θέμα είναι τι μήνυμα θα στείλουμε να αποφασίσουμε, να σας επιβεβαιώσουμε και να αναλάβετε τα καθήκοντά σου επίτροπος. Όλοι θα σκεφτούν τι μήνυμα, όλοι πρέπει να σκεφτούν τι μήνυμα θα στείλουμε. Τι εικόνα στέλνουμε για την Ευρώπη. Λέτε ότι κάνετε λάθη. Όλοι κάνουν, το καταλαβαίνω. Τι προτείνετε σήμερα για να αποφύγουμε την επανάληψή τους. Στην νέα επιτροπή. Θα εμπνευστείτε από τον Βελγικό νόμο του 2005. Θα δημοσιεύσετε διάφορους ε, καταλόγους ε, από Μαυροπίνα και για τα αρπακτικά ταμεία. Θα έχετε όλα τα μέσα, θα κάνετε όλες τις προσπάθειες και έχετε όλες τις εγγυήσεις αμεροληψίας. Για το τελευταίο σημείο. Η κυρία Φόντερ Λάιεν είπε στους πρανσοντολισμούς της ότι ήταν υπέρ μιας τέτοιας προσπάθειας. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που λέτε. Μπορούμε πάντως να το σκεφτούμε. Επίσης είχα πει και στην γραπτή μου παρουσίαση ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου για την ενιαία αγορά να ξαναδούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, που για μένα είναι η βάση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας, ε, ειδικά σε τομείς που έχουν παγκόσμια που εκτίθεται σε παγκόσμιο ανταγωνισμό και που πρέπει παρόλα αυτά η Ευρώπη να προχωρήσει. Θέλω όλοι αυτοί οι τομείς ε, για τους, ε, τις οργανώσεις, τους συνεταιρισμούς, ε, τα ιδρύματα, ε, όλοι αυτοί οι τομείς να ανθίσουν για να μην υπάρχει κατακαιρματισμός εδαφικός ε, στην Ευρώπη και στο εσωτερικό κάποιων χωρών. Και αυτό το βλέπουμε με τον τρόπο που ψηφίζουν οι άνθρωποι που πέφτουν θύματα λαϊκιστών. Επίσης, ε, είμαι υπέρ των νέων που θέλουν να αγωνιστούν και υπέρ μια ε, δίκαιη οικολογική μετάβαση. Θα συνεχίσω να εργάζομαι σε οργανώσει κατά πολέμηση τη στόχια, όπω έκανα μέχρι τώρα, και θα προωθώ και θέματα εσωτερική αγορά παράλληλα. Και τώρα, κυρία Ντεσούτερ, ε, ναι, να ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο με μέλη και των δύο επιτροπών. Πρώτα, ο κύριος Φρανσουά Ξαβιέ Μπελαμή ε, από το ΕΛΚ και την Επιτροπή ΙΤΡΕ, Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Δεν πρέπει εδώ να δημιουργηθεί σύγχυση. Δεν βρισκόμαστε εδώ ε, για να σας κρίνουμε. Θέλουμε να εγγυηθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να λειτουργήσει απρόσκοπτα και αποτελεσματικά. Διαβάσαμε τις απαντήσεις σας, τις γραπτές. Είπατε ότι θα φύγετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα παρεχθείτε μόνο εφόσον υπάρξει οριστική καταδίκη. Ε, ξέρετε ότι η διαδικασία αυτή κρατάει πολλά χρόνια. Ε, η δράση σας ως Επιτρόπου δεν πρόκειται να διακυβευτεί εάν έχετε να διαχειριστείτε μια τέτοια διαδικασία. Έχετε ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο αναλάβει. Ε, και βεβαίω πρόκειται εδώ για τα θέματα περιεχομένου τη ευρωπαϊκή πολιτική. Βεβαίω και σεβόμαστε το τεκμήριο αθότητα, αλλά τίθεται το ερώτημα. Πώ η προσωπική σα κατάσταση δεν θα επηρεάσει τη δράση σα ω Επιτρόπου. Είπατε ότι θα το αποφασίσει αυτό η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό θα αφορά τότε το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπω είναι ένα τρόπο να δημιουργήσετε έτσι ένα πρόβλημα στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη. Το ερώτημα αυτό, για άλλη μια φορά, δεν αποτελεί κρίση για εσά, αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται και το μοιραζόμαστε όλοι. Κύριε Βουλευτά, σα ευχαριστώ. Αυτό που πάτε στο τέλο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα συλλογικό όργανο. Και ο λόγο για τον οποίο ήμουν προσεκτική στην απάντησή μου είναι ότι ε, ό,τι απαντήσω δεσμεύει το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Οποιοδήποτε μέλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να βρεθεί προ μια τέτοιου είδου δυσκολία. Ε, γι' αυτό λοιπόν απάντησα σε δύο φάσει. Ε, μια πολιτική απάντηση που εγώ μπορώ να δεσμευτώ και να πω ότι βεβαίω εφόσον τελικά μου απαγγελθούν κατηγορίε, κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμα, εάν λοιπόν μου απαγγελθούν κατηγορίε όπως το σύνολο των επιτρόπων στον, στους θα μπορούσε να συμβεί αυτό, ενδεχομένως. Ε, στην περίπτωση αυτή λοιπόν, μία είναι η πολιτική απάντηση, να λάβω την ευθύνη μου ανάλογα με την ε, επιμέρους περίσταση και να συζητήσω με την πρόεδρο. Όταν συνεργαζόμουν με τον κύριο Πρόντι, δεν υπήρχε το άρθρο 17 της συνθήκης που έλεγε ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να ζητήσει από έναν επίτροπο να παρετηθεί. Τότε δεν υπήρχε. Το έλεγα και προηγουμένω, ο συνάδελφο από του πράσινου. Αλλάζουν, αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλάζουν οι απαιτήσει. Βρισκόμαστε τώρα προ αυτή τη κατάσταση. Εγώ λάβω αυτή τη δέσμευση ενώπιον σα, αποκοινούμε την κυρία Φόντερ Λάιεν, το συζητήσαμε, το συζητήσαμε και με την νομική υπηρεσία και μετά υπάρχει το αμυγό νομικό κομμάτι. Και εδώ πραγματικά πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα αυτόματος χαρακτήρα παρέτησης δηλαδή πριν από μια καταδίκη. Διότι ε, ο διαχωρισμός ε, των εξουσιών μεταξύ του δικαστικού, του εκτελεστικού τομέα ε, πρέπει να είναι σαφής. Δεν μπορεί να υπάρχει μια ε, διαδικασία δικαστική που να διακυβεύει την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε ότι η ανεξαρτησία είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Μπελαμή, θέλετε να επανέλθετε. Ναι, ακριβώς δεν μιλάμε για κάτι που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Μιλάμε ε, για κάτι που το γνωρίζουμε τώρα, ενώ είστε υποψήφια. Έχω λοιπόν ένα απλό ερώτημα να σας θέσω. Πριν από λίγο καιρό, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είπατε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιλέγει άμεμπτους ανθρώπους. Ε, Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα εμπιστοσύνη ε, στην πολιτική ζωή και γι' αυτό άλλωστε παραιτηθήκατε και στη Γαλλία. Ε, ε, Εμεί δεν προδικάζουμε την ε, ε, καταδίκη σα και την ενοχή σα, αλλά ξέρετε ότι υπήρξαν πίεση σε πολλού συναδέλφου εδώ από αρχηγού κρατών κυβερνήσεων, έτσι ώστε να παραμερίσουμε αυτά τα ερωτηματικά. Μπορεί να μην το γνωρίζετε εσεί. Δεν νομίζετε ότι είναι ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να σα επιτρέψει να δώσετε τι απαντήσει που θα μπορέσουν να εγγυηθούν στους συμπολίτες μας ότι μπορούν να εμπιστευθούν τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξ ολοκλήρου. Νομίζω ότι εσείς θα πάρετε την απόφαση με βάση τη συνείδησή σας. Εγώ σας είπα ό,τι ξέρω, σας έδωσα όλα τα στοιχεία, σας είπα ποια είναι η άποψή μου. Ο καθένας από εσάς θα πάρει την απόφασή του σεβόμενο το σύνολο των αρχών θεμελιών δικαιωμάτων. Να εγγυηθούμε, όπω πολύ σωστά είπατε, την εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα και να εγγυηθούμε βεβαίως και το τεκμήριο αθωότητα. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση. Η κυρία Κούμπουλα Νάτρη, Σοσιαλιστική Ομάδα και από την Επιτροπή Ήτρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις γραπτές απαντήσεις να αναφερθώ σε θέματα βιομηχανικής πολιτικής. Δεν είναι μεταξύ των πέντε προτεραιοτήτων σας, αλλά λέτε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την εξωτερική διάσταση σε συντονισμό με άλλους επιτρόπους. Χόγκαν, Βέσταγερ, Τίμερμανς και άλλοι. Και με άλλους. Είπατε ότι πρέπει οι αρμοδιότητές σας να συνδυαστούν με άλλες και ότι πρέπει να μην υπάρχουν στεγανά στη σύγχρονη εποχή. Ναι, θα ήθελα μερικά παραδείγματα. Ορισμένα παραδείγματα ε, μου αρέσουν, αλλά δημιουργούν ερωτηματικά για τις μικρομεσές ε, και την ψηφιοποίηση. Μία, ένα task force τίθενται και θέματα κινητικότητας ε, στις μεταφορές. Είπατε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι ανοιχτή, αλλά όχι χωρίς μέσα για να αντιμετωπίσει αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Πώς θα συνεργαστείτε με την Επίτροπο Βεστάγκερ, που είπε ότι δεν υπάρχουν ε, επαρκή εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις, χώρες, τις εταιρείες του τρίτου κόσμου που επιδοτούνται. Ευχαριστώ που επανήλθατε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα περιεχομένου. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει περισσότερη συνειδητοποίηση ε, με βάση την κατάσταση όπως αλλάζει στον κόσμο. Διάβασα ένα κείμενο για την κατάσταση στην Κίνα πέρυσι και βλέπω ότι έχει πολύ διαφορετικό τόνο από παλιότερα. Οι εμπορικέ εντάσεις με τις νομές Πολιτείες, ε, νέες χώρες που αναδύονται ω μεγάλε τεχνολογικέ δυνάμει. Όλα αυτά δημιουργούν μια νέα συνειδητοποίηση τη κατάσταση. Να μην κρυβόμαστε. Για πολύ καιρό νομίζαμε ότι σιγά σιγά ο κόσμο θα διαμορφωνόταν όπω θέλουμε εμεί, με κανόνε που να ισχύουν για όλου, με σεβασμό των κανόνων του ΠΟΕ, ότι όλα αυτά ήταν αυτονόητα. Αλλά δεν είναι. Σωστά είπατε. Πρέπει παρόλα αυτά να παραμείνουμε ανοιχτοί γιατί αυτό δημιουργεί ανταγωνισμό, προσελκύει κεφάλαια, προσελκύει ταλαντούχους ανθρώπους. Αλλά, πρώτα απ' όλα, θα έχουμε αυτό το νέο μηχανισμό για έλεγχο των εξωτερικών επενδύσεων. Αν υπάρξει εξωτερική επένδυση, για παράδειγμα μόνο και μόνο για να μας κλέψει τεχνολογίες, δεν θα το αφήσουμε. Για παράδειγμα, στη Γερμανία γίνονται ορισμένε εξαγορέ επιχειρήσεων μόνο και μόνο για να κλέψουν τεχνολογία. Αυτό δεν θα πρέπει να το επιτρέπουμε. Άλλε όμω θα πρέπει να τι επιτρέπουμε. Είμαι πεπισμένη ότι η ανταγωνιστικότητα. Συγγνώμη, ο ανταγωνισμό βοηθάει την ανταγωνιστικότητα. Βεβαίω πρέπει να έχουμε κανόνε για τον ανταγωνισμό, αλλά να του προσαρμόσουμε σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Όλα αυτά τα μεγάλη διάσταση ε, εγχειρήματα που επιτρέπουν σε συγκεκριμένο τομέα όπως για παράδειγμα για τις μπαταρίες, επιτρέπουν να συνδυάσουμε πόρους χωρίς να υπαγόμεθα στους κλασικούς κανόνες ανταγωνισμού. Διότι ξέρετε ότι παλιά οι απαγορεύσεις για, τον, για τις επιδοτήσεις ήταν για να παρεμποδίσουν τις μεγάλες χώρες να βοηθήσουν πολύ περισσότερο τις εταιρείε τους από τις μικρές χώρες. Νομίζω ότι δεν έχουμε διαφορά αντιλήψεων ε, μεταξύ μας σε αυτό το θέμα. Συνοματική ερώτηση. Η βιομηχανική στρατηγική είναι ευθύνη σας. Αλλά είναι τμήμα του μεγαλύτερου οικοσυστήματος δημιουργίας ε, δυνατοτήτων. Αλλά δεν μπορούμε να το δούμε ξεχωριστά από τους ε, κανόνες ανταγωνισμού, γιατί θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Και όλοι θέλουμε να στηρίξουμε τις ε, πρωτοπόρες ευρωπαϊκές εταιρείες, χωρίς όμως να περιορίσουμε τις ε, επιλογές για τον καταναλωτή. Πώς θα βοηθήσουμε λοιπόν σε ένα νέο σύγχρονο κόσμο αυτές τις πρωτοπόρες ευρωπαϊκές εταιρείες. Κοιτάξτε. Τι επιτρέπει ως συγχωνεύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγκρίνει το 95-96% των ε, συγχωνεύσεων που τις υποβάλλονται. Επίσης, έχουμε τέτοιες καλές ευρωπαϊκές εταιρείες, πρωτοπόρες. Για το 5G, για παράδειγμα. Η Nokia και η Ericsson ηγούνται της εισαγωγής των 5G. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι έχουμε χάσει αυτόν τον αγώνα. Ορισμένε επιχειρήσει μα ηγούνται διαφόρων κλάδων. Σε άλλου κλάδου υπολοιπόμεθα. Γι' αυτό επιμένω στην τεχνολογία, όπω είπα και στην εισαγωγή μου. Μόνο αν διατηρήσουμε τι άριστε εταιρείε θα βοηθήσουμε την οικονομία μα. Η καλύτερη προστασία, η καλύτερη ασπίδα είναι να είσαι ο καλύτερος, να έχει καλά πανεπιστήμια, να έχει καλού νέου ερευνητέ που να μην φεύγουν από την Ευρώπη, να έχουν προοπτικέ μέλλοντο να είμαστε ισχυροί. Οι κανόνες του ανταγωνισμού μπορούν να βοηθήσουν, να συνοδεύσουν για αυτά τα μεγάλα εγχειρήματα ευρωπαϊκής διάστασης, αλλά η καλύτερη προστασία είναι η αριστεία. Πρέπει να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας ε, που ηγούνται κάποιου κλάδου να ηγηθούν ακόμη περισσότερο. κυρία από και την Επιτροπή Ευχαριστώ. Θα μιλήσω τσέχικα. Επίτροπε, υποψήφια επίτροπε, αγαπητή Σιλβή, πάρα πολλές ερωτήσεις τις βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τη συζήτηση και σέβομαι τη γαλλική εσωτερική πολιτική, αλλά με πάνω αυτό στο χαρτοφυλάκιό σα. Αντίθετα από πολλού συναδέλφου, εγώ διάβασα πολύ εντελεχώ τι γραπτέ σα απαντήσει και χαίρομαι για όλα όσα λέτε για την προστασία ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι 24 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ήταν προτεραιότητα και του τελευταίου Επιτρόπου ε, με πολλές ε, πρωτοβουλίες, αλλά δεν υλοποιήθηκαν όλοι, όλες τις πρωτοβουλίες. Στις γραπτές ε, απαντήσεις είπατε ότι πρέπει να μειωθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να αντιμετωπίσετε τις καθυστερημένες πληρωμές. Σωστά είναι αυτά και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Μία ερώτηση τώρα. Έχετε μια σαφή ιδέα για το πώς θα τα εφαρμόσετε όλα αυτά, πώς θα τα κάνετε πραγματικότητα Πώς θα εφαρμόσετε και θα παρακολουθήσετε την πρωτοβουλία στη νέα στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα χρησιμοποιήσετε το ευρωπαϊκό εξάμεινο και ανέπω, ναι, πώς, κυρία Γκουλάχ. Ευχαριστώ. όταν έχουμε 24 εκατομμύρια επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ άριθμες. Ε, υπάρχουν μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις με τεράστια δημιουργικότητα. Σε ορισμένε ε, χώρες έχουμε νεοφύης επιχειρήσεις, αλλού μεγαλύτερες. Θέλουμε να δουλέψουμε σε πολλά επίπεδα. Όπως είπα και στην πρώτη μου εισαγωγή, θέλω να είμαι όσο πιο ρεαλίστρια γίνεται. Κάθε φορά που είχα συναντήσεις με επικεφαλής επιχειρήσεων, ε, δεν μου ζητούσαν φοβερές στρατηγικές οι διευθυντέ αυτοί. Θέλουν συγκεκριμένα πράγματα. Θα πρέπει η οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές να εφαρμοστεί πάρα αυτά και αυτή είναι αρμοδιότητα του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχουν και θέματα χρηματοδότησης. Το είπατε κι εσείς. Κάποια ταμεία υπάρχουν για να επεκταθούν οι επιχειρήσεις για να μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις. Θα πρέπει να τα προωθήσουμε αυτά τα εργαλεία. Στο Investing You, στο νέο πρόγραμμα, αν υιοθετηθεί το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί το θέλει αυτό η Επιτροπή και ελπίζω εδώ να βοηθήσει και το Βουνούλιο, έχουμε ταμεία και κονδύλια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μία ιδέα ήταν να έχουμε ένα πεσταλμένο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να είναι ο συνομιλητής τους και να με βοηθάει σε σχέση με τις μικρομεσαίες μέχρι τώρα. Ο επίτροπο το έκανε αυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει κάποιο να δουλεύει 100% εκεί. Στο ψηφιακό τομέα ε, υπάρχει η πράξη για τι ψηφιακέ ε, υπηρεσίε. Υπάρχει και εκεί ένα κομμάτι για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Σα φαίνονται κατακαιρματισμένα όλα αυτά, αλλά στην πραγματικότητα ε, καλύπτουμε όλε τι ανάγκε που έχουν οι διευθυντέ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι διοκτήτε του. Υπάρχουν και πράγματα που αφορούν άλλου συναδέλφου. Ω ο επίτροπο που είναι υπεύθυνο για το περιβάλλον ή τη θέση απασχόληση, θα παίξουν και αυτοί κάποιο ρόλο για το θέμα αυτό. Συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ για τις λεπτομερείς σας απαντήσεις. Όπως είπατε και στις γραπτές σας απαντήσεις, στην αρχική φάση προετοιμασίας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όταν αξιολογούμε την επίπτωση, είναι σημαντικό να λάβουμε επίπτωση κάθε, της κάθε πολιτικής πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς θα αποφύγουμε την νομοθεσία η οποία είναι πάρα πολύ επαχθής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυξάνει πολύ το γραφειοκρατικό άχθος. Είπατε ότι πρέπει να συνεργαστούν διάφορες γενικές διευθύνσεις ε, και εσείς με διαφόρους συναδέλφους σας στην Κομισιόν. Πώς θα διαμορφωθεί αυτή η συνεργασία με τον Μάρος Σεύκοβιτς, που είναι επίτροπος, ε, που έχει επίσης αρμοδιότητες που εφάπτονται με τις δικές σας. Πώς θα μειώσετε το γραφειοκρατικό άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεργασία με τους συναδέλφους σας. Η κυρία Γκουλά, ευχαριστώ. Δεν είχα την ευκαιρία μέχρι στιγμής να αναφερθώ τον κύριο Σεύκοβιτς που έχει βαρύ καθήκον να έχουμε καλύτερη νομοθεσία. Αυτή είναι η αρμοδιότητά του. Θα πρέπει να έχουμε τον εξή αυτοματισμό. Όταν ετοιμάζουμε ένα κείμενο, θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι επίπτωση θα έχει στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Το έκανε και η προηγούμενη ε, Κομισιόν, αλλά αν το σκεφτούμε περισσότερο, θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Επίση, θα πρέπει να συζητήσουμε μαζί όταν είμαστε στην αρχική φάση της νομοθεσίας. Άλλοι σε Αλλιώς σκεφτόμαστε στο πρωτογενές δίκαιο και όταν ε, υιοθετούμε κατεξιοδότηση και πράξεις, ας πούμε. Εγώ τα έχω ζήσει όλα αυτά. Δεν θα σας υποσχεθώ βέβαια ότι μια νυχτή όλα θα γίνουν καλύτερα, αλλά ξέρω πολύ καλά τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βλέπω ότι πολλά αφεντικά δυσκολεύονται, έχουν δύσκολη καθημερινότητα. Πολλέ όμω θέσει απασχόληση εξαρτώνται από την ευμερία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά θα, θα τι έχουμε πάντα στο μυαλό μα. Ευχαριστώ κυρία Σόντροφα τώρα ε, από το ΕΛΚ και την Επιτροπή Πολιτισμού. Ευχαριστώ πολύ κυρία υποψήφια Επίτροπε. Στις γραπτές σας απαντήσεις μας διασφαλίσετε ότι το πρόγραμμα Media, ο τομέας των οπτικοκουστικών θα είναι από τις μεγάλες σας προτεραιότητες λόγω της μοναδικής του σημασίας ε, σε πολιτιστικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Από αυτά που διάβασα όμως, θεωρώ ότι ο κλάδος αυτός ε, ουσιαστικά το βλέπετε υπό το πρίσμα της ψηφιακής ε, τεχνολογίας και της εσωτερικής αγοράς. Δεν βλέπω να υπάρχει ιδιαίτερη κατανόηση σε ό,τι αφορά τον πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο του τομέα αυτού. ποιο είναι το δικό σας όραμα για την πολιτική ε, στον οπτικοκουστικό τομέα και στον τομέα των μέσων ενημέρωσης. Πώς ε, ταιριάζουν στο όραμα αυτά τα στοιχεία ε, το, στο όραμά σας και πώς θα εξασφαλίσετε ότι θα υπάρχει απόλυτη προστασία και αναγνώριση της, του πολιτισμού στη δράση σας. Κυρία Γκουλάρ, ε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να επανέλθω στο θέμα αυτό διότι ακούσατε αυτά που σας είπε η Μαρία Γκαμπριέλε όταν ήρθε εδώ ε, και εδώ θα πρέπει να συνεργαστούμε. Δεν νομίζω να υπάρχει εδώ κάποια αντίθεση και αντιπαράθεση. Η σημασία του πολιτισμού, η υποστήριξη της δημιουργίας, το να βοηθήσουμε όλα τα επαγγέλματα δημιουργών, είτε δημιουργούν βιντεοπαιχνίδια, είτε κινηματογραφικές ταινίες που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε άλλα άλλους τύπους περιεχομένων. Ε, είναι ένας από τους θησαυρούς της Ευρώπης. Όλοι αυτοί οι δημιουργοί που συνεισφέρουν ε, στο να προστατευτεί η ποικιλομορφία της Ευρώπης και να λάμψει η Ευρώπη ανά τον κόσμο. Ε, και υπάρχει αυτή η ιδέα ε, συγκεκριμένων υποχρεώσεων για πολιτιστική, πολιτιστική ποικιλομορφία. Εφόσον υπάρχουν υποχρεώσεις ό,τι αφορά ε, την διανομή, πρέπει να υπάρχουν υποχρεώσει και για το τομέα τη δημιουργία. Δηλαδή, κάποιοι δημιουργούν κάποια πράγματα και κανεί δεν έχει πρόσβαση σε αυτά. Ε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Αυτή είναι μια στι πρώτε προτεραιότητέ μου, λοιπόν. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω το είπαμε και προηγουμένω για τι μεγάλε πλατφόρμες, για να μπορέσει η δημιουργία στην Ευρώπη ε, να μην σταματήσει, θα πρέπει να μειώσουμε την εξουσία που έχουν τις μεγάλες πλατφόρμες στην αγορά και τον τρόπο με τον οποίο εγκαθίστανται στον τομέα των ιδεών, της ε, διανομής, ε, του πολιτικού τομέα γενικότερα. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε σωστά μια οδηγία η οποία έχει ήδη εγκριθεί. Τέλος υπάρχει το θέμα της οικονομικής υποστήριξης μέσω του προγράμματος Media που δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Αυτό οδηγεί στην παραγωγή ταινιών που ε, βραβεύονται, που ε, προβάλλονται στο σύνολο του ευρωπαϊκού εδάφους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν και κάποιες εργασίες, ε, τώρα τα ανακαλύπτω αυτά ομολογώ, ε, εργασίες για τον υποτιτλισμό των ταινίων. Πώς μπορούμε να έχουμε μια βάση δεδομένου με τους υπότιτλους. Πώς μπορούμε όλες, να, να, να βοηθήσουμε έτσι ώστε όλη αυτή η πολιτική δημιουργία να μπορεί να περνάει πιο εύκολα τα σύνορα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα του πολιτισμού. Ε, θα πρέπει η διάβλη διανομής όμως του πολιτισμού να είναι ισχυροί, να προστατεύονται και έτσι θα εγγυηθούμε την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρώπης. Κάποια δεύτερη ερώτηση. Ναι, βεβαίως. Θα ήθελα να συμπληρώσω το ερώτημά μου, διότι δεν κρύβω ότι είμαι κάπως ε, απογοητευμένη. Ε, ε, μας επαναλάβετε το τι έχουμε κάνει. Μας επαναλάβετε τα προβλήματα. Τα γνωρίζουμε τα προβλήματα έχουμε τις νέες ε, μορφές τεχνολογιών, την ε, τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να προστατεύσουμε τον κλάδο, να τον αναπτύξουμε όμως εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε, ποιες είναι οι δράσεις που θα αναλάβετε σε νομοθετικό επίπεδο, σε προγραμματικό επίπεδο, ε, ποιος θα είναι ο προπολογισμός. Θέλουμε να ακούσουμε κάτι συγκεκριμένο για τη δική σας προσέγγιση. Τι θέλετε να βελτιώσετε. Σας ευχαριστώ που επανέρχεστε. Ναι, αυτός είναι πάντο κίνδυνος όταν βλέπουμε τα θέματα ένα προς ένα. Πριν μίλησα ε, για την ε, νομοθετική πράξη και τις ψηφιακές υπηρεσίες, ε, Τεχνητή νοημοσύνη επίση δεν το συζητήσαμε τώρα, αλλά τα ανέφερα στι τελευταίε μου απαντήσει. Υπάρχουν πολιτικές που φαίνονται να μην συνδέονται με τα ζητήματα πολιτισμού. όμως ένα μέρος της δουλειά μα, τη δουλειά θα πρέπει να γίνει. Και αυτό το έχουμε μπροστά μα, όχι πίσω μα ε, σε ό,τι αφορά την νομοθετική πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα είναι αφενός να προστατεύσουμε κάποιες αρχές που έχουν να κάνουν με τις οδηγίες που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή και αφετέρου να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα περιεχόμενα, ε, να εργαστούμε πάνω στο θέμα των, των πλατφορμών και να πλαισιώσουμε καλύτερα την εξουσία τους. Ε, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη που θα οδηγήσει ε, σε κάποια αποτελέσματα σε ηθικό επίπεδο και σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί ε, και στον τομέα του πολιτισμού. Είναι άλλη μια πόρτα εισόδου αυτή. Μου λέτε και τον προπολογισμό. Ε, ξέρετε, δεν του καθορίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνη τη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει προτάσει και από εκεί πέρα τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι πολύ φιλόδοξε προτάσει αυτέ. Βοηθήστε μα λοιπόν στη μάχη αυτή, έτσι ώστε οι προπολογισμοί αυτοί να μπορέσουμε να του υπερασπιστούμε. Ε... Ευχαριστώ. Κυρία Σοσιαλίστρια από την ΜΜΚΟΜ. Ευχαριστώ. Κυρία Γκουλάρ, ακούσαμε και διαβάσαμε τα σχόλια για την ακυρότητά σα. Ω ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών σημειώνουμε τι απαντήσει σα. Ωστόσο, θα παρακολουθήσουμε την εργασία σα και την ακυρότητά σα αν βεβαιωθείτε. Αλλά νομίζω ότι είναι θέμα τη κυρία Φοντελάιν τώρα να κάνει μια σαφή δήλωση για να βελτιωθεί ο κώδικα διοντολογία. Ερώτηση. Κοινωνική αγορά αναφέρεται επανειλημμένα στις γραπτές απαντήσεις σας. Αλλά δεν βλέπω καλά τον σύνδεσμο μεταξύ κοινωνικών θεμάτων και ενία αγοράς. Το βλέπω σε διάφορες δηλώσεις συναδέλφων σας, αλλά όχι στις δικές σας. Πώς η ενιαία αγορά θα βοηθήσει να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. Ευχαριστώ κύριε Γκουλάου. Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Μερικά από όσα λέω έχουν να κάνουν με τη δράση του συνόλου των επιτρόπων. Τώρα θα επικεντρώσω στις δικές μου αρμοδιότητες. Το είπα και στον κύριο Μπομπά προηγουμένως. Πρέπει να εμείνουμε σε μια κοινωνική και αλληλέγγυα ε, οικονομία, όπου κάποιες επιχειρήσεις ε, που ασχολούνται με αυτούς τους τομείς να είναι η κύρια προτεραιότητά μας. Είναι επιχειρήσεις που ασχολούνται σε διάφορες περιοχές με καινοτόμους ε, τρόπους για να σεβαστούμε και τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς αλλά και από πλευρά συμπεριφοράς συμπεριφορά των επιχειρήσεων δηλαδή ο συνεργατικός τομέας τα διάφορα ιδρύματα οι διάφορες συνεργατικές επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλλουν στην παροχή υπηρεσιών τοπικά. Μπορούν να βρουν νέες λύσεις για την κινητικότητα που θα βοηθήσουν το κλίμα. Μπορούν να συμβάλλουν για να υπάρξει περισσότερη αλληλεγγύη, έναντι των ηλικιωμένων που είναι όλο και περισσότεροι. Κάποια άτομα που είναι κάπως στο περιθώριο μπορεί να βοηθηθούν να επανέλθουν στην οικονομική δραστηριότητα. Είναι σημαντικό τμήμα της ε, εργασία μου. Επίση, ορισμένα θέματα που έχουν να κάνουν με την οδηγία για τι υπηρεσίε. Ξέρετε ότι το πρόβλημα που έχουμε ορισμένε φορέ είναι ότι όταν τα άτομα του προσωπικού, δηλαδή μια επιχείρηση, θέλουν να ε, περάσουν τα σύνορα, αντιμετωπίζουν πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια. Μου έχει επισημανθεί επανειλημμένα. Εκεί θα συνεργαστώ με τον Νικολά Σμιτ, γιατί είναι ένα τμήμα, ε, είναι ένα μέρος θέμα υπηρεσιών και ένα θέμα κοινωνικής αγοράς για να έχουμε συγκεκριμένε λύσεις για τα άτομα που θέλουν να εργάζονται σε δύο διαφορετικές χώρες σεβόμενοι πάντα τους κοινωνικούς κανόνες. Παρακαλώ, σημαντική ερώτηση. Ναι, για την οδηγία της υπηρεσία. Θέλουμε συγκεκριμένα τη θέση σα. Είπατε ότι δεν θα την ξανανοίξετε. Αλλά θα σεβαστείτε πλήρως τι θεμελιώδει αρχέ αυτή τη οδηγία. ή όχι η θεμελιώδης αρχή να εφαρμόζεται η θεμελιώδη αρχη να εφαρμοζεται η αρχη της χώρας προορισμού. Γιατί έτσι θα δημιουργήσουμε περισσότερη συνοχή. Συγγνώμη, της χώρας προέλευση. Δεν θεωρείτε ότι είναι θεμελιώδε. Κοιτάξτε, δεν θέλουμε να ξανακάνουμε όλες τις αντιπαραθέσεις που έχουν γίνει. Θα πάρω τα κείμενα όπως είναι και τις αρχές των συνθήκων. Να μην έχετε καμία ανησυχία και αμφιβολία. Δεν θα ξανακάνουμε μία μάχη που έχει ήδη γίνει γιατί αυτό θα καταστρέψει την εμπιστοσύνη αντί να οικοδομήσει περισσότερη εμπιστοσύνη που θα μας δημιουργήσει να προχωρήσουμε. Η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι θεμελιώδης γιατί όλοι οι άλλοι τομείς είτε είναι η βιομηχανία είτε η γεωργία, περιλαμβάνουν όλο και περισσότερες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, μέσω του νομοθετήματος για τις ψηφιακές υπηρεσίες μπορούμε να λάβουμε κάποια μέτρα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των εργαζομένων πλατφόρμες. Αυτά τα θέματα δεν ήταν πρώτη προτεραιότητα όταν ανακρίθησαν αυτά τα κείμενα λεπτών των αρχών, είναι σαφές. Και για τα άλλα, ούτως ή άλλως, εάν με εμπιστευτείτε, θα τα συζητήσουμε Ξέρετε ότι η Επιτροπή κάνει προτάσεις και η εργασία που είχε κάνει η κυρία Γκεπάρτ και άλλοι στο παρελθόν θα συνεχιστεί. Επί των αρχών θέλω να είμαι σαφής. Αλλά ε, οι διαδικασίες, ο εξυγχρονισμός θα συνεχιστούν. Τελευταία ερώτηση στο δεύτερο γύρο, κυρία Βάης, από το EPP Ήτρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, έχω την τιμή να θέτω την τελευταία ερώτηση σήμερα θα, να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα τα δανέζικα, αν μου επιτρέπετε. Εμείς θέλουμε πολύ ψηλά πρότυπα όσοι έχουν δημόσια λειτουργήματα, όσοι είναι υπουργοί, όσοι είναι στην κυβέρνηση. Ως υπουργό είχατε ένα από τα υψηλότερα πόστα στη Γαλλία. Ε, επιλέξατε να παρτηθείτε λόγω μιας ε, υπόθεσης η οποία τρέχει ακόμα, η οποία ερευνάται ακόμα στη Γαλλία και τώρα είσαστε υποψήφια για ένα από τα υψηλότερα πόστα, τη σημαντικότερε θέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο ΕΛΚ πιστεύουμε ότι τα ίδια υψηλά πρότυπα θα πρέπει να ισχύουν για όσους κατέχουν υψηλά αξιώματα σε εθνικό επίπεδο με αυτού που κατέχουν υψηλά αξιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας δώσω μια τελευταία ευκαιρία να μας εξηγήσετε γιατί θα πρέπει να δεχτούμε χαμηλότερα πρότυπα από αυτού που επιδιώκουν ένα δημόσιο αξίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτούς που έχουν κάποιο δημόσιο αξίωμα στη Γαλλία. Κύριε Σας ευχαριστώ που επανέρχεστε ακόμα μια φορά σε αυτό το θέμα. Θα επαναλάβω αυτά που έχω ήδη εξηγήσει. Παρουσιάσατε τα πράγματα ω εξή. Ότι ο νόμο γαλλική δημοκρατία θα πρέπει να ισχύει παντού. Αυτό είναι επικίνδυνο, πιστεύω. Εγώ δεν ισχυρίστηκα κάτι τέτοιο. Μου θέσατε ερωτήσει για το τι έχω κάνει. Έχω δεσμευτεί πολιτικά ενώπιό σα, αφού συζήτησα με την κυρία Φόντερ Λάιεν. Η κυρία Φόντερ Λάιεν και εγώ φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι μπορώ να αναλάβω μια πολιτική δέσμευση, αλλά δεν υπάρχει νομικός αυτοματισμός λόγω των διαφορετικών νομικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν ξέρω το δανέζικο δίκαιο, το ομολογώ. Δεν ξέρω το δίκαιο στα περισσότερα κράτη-μέλη ό,τι αφορά την ποινική διαδικασία. Θα πρέπει όλοι οι επίτροποι να αντιμετωπίζονται ισότιμα και όλοι οι επίτροποι να μην υφίσταται διακρίσει. Να μην υπάρχει καμία απόπειρα αποσταθεροποίηση τη Κομισιόν μέσω εν εξελίξη νομικών διαδικασιών εις βάρος ενός ε, επιτρόπου ε, και όταν κάτι δεν είναι ξεκάθαρο να μην γίνεται τίποτα αυτόματα. Όταν λέω ότι δεν πρέπει να γίνεται κάτι αυτόματα, τι σημαίνει. Ότι νομικά δεν βγάζουμε συμπεράσματα πριν την ώρα μας, αλλά την πολιτική δέσμευση δεν μπορούμε να την ε, εμποδίσουμε. Μπορεί να υπάρχει πολιτική δέσμευση, και μπορεί να υπάρχει και πολιτική ε, ευθύνη. Επίσης, ε, ίσως άκουσα κάτι που δεν ξέρω είναι σωστό. Δεν το άκουσα καλά. Ποτέ δεν μου απαγγέλθηκε κατηγορία. Ποτέ. Εγώ παίρνω τις αποφάσεις μου με τα λόγου γνώσεως. Εσείς μιλήσετε για την ακαιρεότητα των πολιτικών. Είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει όμως και κάποια άλλη βασική αρχή που είναι το τεκμήριο αθωότητας. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση. Είπα ότι πρέπει να παρετηθείτε λόγω μιας υπόθεσης η οποία ακόμα ερευνάτε. Από την απάντησή σας συλλέγω ότι δεν θα κάνετε τίποτα και ότι δεν αμφιβάλλετε ότι θα πρέπει τα ίδια πρότυπα να ισχύουν για τους ε, υπουργούς, ας πούμε, στη Γαλλία με τους επιτρόπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχω άλλη ερώτηση να σας προσθέσω και κάτι άλλο. Υπάρχει μια αμφισημία για την κατάσταση στη Γαλλία. Στη Γαλλία δεν υπάρχει κάποιος κανόνας. Υπάρχει το εθνικό δίκαιο. Όταν παραιτήθηκα από Υπουργό Άμυνα, ήταν μια πολύ ειδική στιγμή μετά την εκλογή του Προέδρου τη Δημοκρατία και ήταν μια πολύ διαφορετική πολιτική συγκυρία. Δεν νομίζω ότι πρέπει να λένε ότι υπάρχουν διπλά μέτρα και σταθμά. Ζούμε στην Ευρώπη, υπάρχει επικουρικότητα, μπορεί να υπάρχει μια χώρα η οποία αποφασίζει να πάει πιο μακριά σε κάποιου τομεί. Το μόνο που μπορώ να σα πω είναι ότι το συζήτησα με την κυρία Φόντερ Λάιον, είναι η πρόεδρο αυτή τη επιτροπή και μάλιστα είναι και από την πολιτική σα ομάδα. Μπορείτε να την εμπιστευτείτε ότι θα είναι πάρα πολύ αυστηρή. Εγώ από μόνη μου δεν μπορώ να προβλέψω κάτι που δεν το, προβλέψουν, δεν το προβλέπουν οι συνθήκες. Και οι νομικοί της ε, Κομισιόν θεωρούν ότι αν προκύψει αυτός ο αυτοματισμός θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ την κυρία Γκουλάρα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ο δεύτερος γύρος ερωτήσεων από τις Επιτροπές. Καλό τώρα ε, την ε, υποψήφια Επίτροπο ε, να κάνει μια τελευταία δήλωση, όχι πάνω από 5 λεπτά παρακαλώ. Κυρία Γκουλάρ, ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες ε, Πρόεδροι και εξωτιμοί κύριοι Ευρωβουλευτές. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων. Υπήρξε μεγάλη, υπήρξε ένα πνεύμα ευγένεια. Ε, προσπάθησα να απαντήσω. Συζητήσαμε πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έμαθα, σας γνώρισα καλύτερα. Μπορούσαμε να πούμε και να συζητήσουμε σε βάθος κάποια από τα ζητήματα. Είναι θεμητά τα ερωτήματά σας. Απάντησα με βάση τις επιπιθήσεις μου. Δεν λέω ε, ότι γνωρίζω τα πάντα για όλα τα ζητήματα τα οποία μου έχουν ε, ανατεθεί. Δεν νομίζω όμως ότι και όλοι οι επίτροποι ε, γνωρίζουν όλα τα θέματα που έχουν αναλάβει πλήρως. Σιγά σιγά θα μάθουμε. Σέβομαι ιδιαίτερα πάντως αυτή τη διαδικασία πρέπει να πω συχνά ακούω να λέγεται ότι η Ευρώπη πάσχει από δημοκρατικό έλλειμμα. Ακούμε πολύ συχνά αυτή την έκφραση. Είμαι εδώ όμω ε, σήμερα για δεύτερη φορά ενώπιον σα και δεν νομίζω να υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα. Υπάρχει ένα σοβαρό, αυστηρό έλεγχο ε, των ε, υποψήφιων επιτρόπων και αυτό είναι καλό. Ελπίζω να αξιολογήσετε ένα πρόσωπο, ένα άτομο, τη σταδιοδρομία του, τη διαδρομή του με ό,τι έχω κάνει εδώ και 30 χρόνια. Ε, έχω ζήσει συναρπαστικές στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας. Όλα αυτά που συνέβησαν το 1989, πριν από 30 χρόνια, όταν ξεκίνησα την καριέρα μου στην γαλλική διπλωματία και που συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις για την, για την επανένωση της επανένωση της Γερμανίας και στη συνέχεια με τη διεύρυνση υπό τον Ρωμάνο, Φρό, τον Ρωμάνο Πρόντι. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο χρονικό διάστημα. Όλες αυτές οι αλλαγές ε, οι παγκόσμιες που έχουμε μπροστά μας δίνουν στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση περισσότερο οποιαδήποτε άλλη στιγμή έναν λόγο ύπαρξης. Περισσότερο οποιαδήποτε άλλη στιγμή πρέπει να είμαστε ενωμένοι, ε, πρέπει να ενώσουμε τις οικονομικές, ε, τις πολιτιστικές μας δυνάμεις. Είναι μια παλιά ήπειρος η Ευρώπη, αλλά έχει πολλά ακόμα να προσφέρει στον κόσμο. Μπορεί να είναι μια μέση οδός ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες δυνάμεις που αυτή τη στιγμή ε, είναι, βρίσκονται αντιμέτωπε. Θέλω λοιπόν να, να κρίνετε, με κρίνετε ω άτομο, ω διαδρομή. Είπατε κύριε Μπελαμίου ότι δεν είστε εδώ για να κρίνετε. Αξιολογείτε όμω. Ε, προσωπικά θεωρώ ότι είναι συναρπαστικό αυτό το χαρτοφυλάκιο, αυτή η θητεία που μου προτείνετε. Ελπίζω να μου δώσετε την ευκαιρία να ασκήσω τα καθήκοντά μου μαζί με την κυρία Φόντερ Λάιν. Είναι μεγάλη η ομάδα μα. Ε, δεν μπορούσα να μιλήσω για όλου. Ε, είμαστε μία ομάδα, έτσι. Εγώ είμαι ένα μέλος τη ομάδα αυτής. Έχετε αξιολογήσει του περισσότερου από αυτούς. Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τη διαδρομή μου, την δέσμευσή μου και ε, εφόσον, όταν θα τα ξαναπούμε, ελπίζω να τα πούμε υπό καλές συνθήκες. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την διαδικασία ε, άσκησης ε, δημοκρατίας διασυνοριακής. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ κυρία Γκουλάρ για την δήλωσή σας, για τις απαντήσεις που δώσατε στα μέλη και των δύο επιτροπών. Εκ μέρους της Επιτροπής ΙΜΚΟ, καλώς ορίζω όλα τα μέλη. Έχουμε ακόμα κάποιες ανακοινώσεις να κάνουμε. Σας ευχαριστώ όλους όσους ήρθατε. Και θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Βαλεάν για να κλείσει τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ και εγώ όλους όσους συμμετείχατε σε αυτή την προσπάθεια. Τώρα θα πρέπει να αξιολογήσουμε αυτή την ακρόαση, συνάδελφοι. Αυτό θα γίνει και κλεισμένο των θυρών από τους συντονιστές και η συνεδρίαση θα γίνει εδώ στις 12.30.